Okay, if everybody would sit down. Καθίστε παρακαλώ όλοι. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 10 της σήμερα της διατάξης, ο οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντίσεμπλουμ. έρχεται, παίρνει το βάπτισμα του πυρός, διότι είναι δύσκολη η καιρή αυτή. Έτσι μπορούμε να το περιγράψουμε. Η κατάσταση στην Κύπρο, που παρακολουθήσαμε πώς εξελίχθηκε το Σαββατοκυριακό, είδαμε τις αντιδράσεις στο πακέτο που είχε συμφωνηθεί και η αντίδραση δημιούργησε πολλές ανησυχίες και για μένα και για άλλα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαι βέβαιο ότι πρέπει να καλυφθούν και άλλα θέματα σήμερα, πέραν αυτού αλλά θα ήθελα στην εισαγωγική του παρουσίαση να μας πει πότε διαπίστωσε ότι θα υπήρχαν προβλήματα με το συμπεφωνημένο πακέτο. Ίσως μπορεί να μας περιγράψει αναδρομικά πως έφτασε η κατάσταση εκεί που έφτασε. Αναφέρονται πολλά στον τύπο. Ίσως μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες χωρίς να ξεκινήσουμε κάποιο κυνήγι μαγισσών. Έχω μία ερώτηση. Γιατί όταν βγήκαν με κάποιο τελικό πακέτο γιατί δεν δείχτηκε κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία στην δήλωση. Σε εκείνη τη φάση να επισημανθεί ότι για πολλούς θα φαινόταν ότι η συμφωνία θα είχε παραβιαστεί την εμπιστοσύνη, την εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ. Ξέρω ότι μπορεί να το ξεπεράσει κανείς να πει ότι είναι ένας φόρος, μια εισφορά, φόρος ε, πλούτου αν θέλετε, αλλά αναφυσβήτητα στο μυαλό πολλών πολιτών, όπω ξέρουν οι Ευρωβουλευτέ, δημιουργήθηκαν πάρα πολλέ ανησυχίε. Τι είναι αυτό, καινούριο εργαλείο στην εργαλειοθήκη, ε, τι μπορούμε να περιμένουμε, υπάρχει ασφάλεια. Και ίσω να μα. Ίσως με καλύτερη εξήγηση για το πακέτο Ίσως να καθησύχαζαν περισσότερο αυτοί που θα άκουγαν το μέτρο εκ των προτέρων, αντί να περιμένουν μια δεύτερη δήλωση που ε, ακολούθησε και ίσως να ήταν ε, πολύ σύντομη σε μια προσπάθεια φυσυχασμού των δημιουργηθισών ανησυχιών. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω αυτή να είναι μια πρώτη από πολλές ε, ανταλλαγές απόψεων και ίσως στο μέλλον να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες για τις επόμενες συναντήσεις. Ακολουθούμε την εξή προσέγγιση. 10 λεπτά για μια παρουσίαση δεν θα είναι αρκετό ο χρόνο για να καλύψετε όσα θέλετε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και μετά θα πάμε σε πεντά λεπτά για ερωταπαντήσει ε, και απευθύνω εκ των προτέρων έκκληση προ τα μέλη. Παρακαλώ, παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε σύντομοι σε ερωτήσει, ούτω ώστε να υπάρχει χρόνο για να απαντήσει ο Υπουργό. Και αν είστε αρκετά σύντομοι και απαντήσει αρκετά γρήγορα, τότε μπορείτε να δευτερολογήσετε και πιθανότατα έτσι να το αποσπάσετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Ε, thank you, Madam Chair. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω σταθεί βοηθός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1993. Ήταν η πρώτη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου. Τότε δεν υπήρχε αυτό το κτίριο, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν πολύ διαφορετικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που επιστρέφω βέβαια με μια τελείως διαφορετική ιδιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για τη μόνιμη συμμετοχή της στη συζήτηση των οικονομικών και νομισματικών θεμάτων. Ενώπιον σας σήμερα Έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι η Επιτροπή σας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νομοθεσία στα θέματα αυτά και παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν αυτή την ευκαιρία και τις μελλοντικέ ευκαιρίες για να έχουμε ανταλλαγέ απόψεων και να χρησιμοποιήσω και την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής αυτής. Η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις η εστίασή μα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίω η αντιμετώπιση κρίσεων. Όπω ξέρετε αυτή τη στιγμή οι εξελίξει στην, στην Κύπρο βρίσκονται στο προσκήνιο και του δικού μου και του δικού σα μυαλού φαντάζομαι. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωομάδα πέτυχε μια πολιτική συμφωνία με τι πολι... με για τα κύρια σημεία ενό προγράμματο προσαρμογή ύψου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2016. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό δημοσιονομική εξυγίανση, διαφορετικές αλλαγές, ιδιωτικοποίησεις και θα επέτρεπε το κυπριακό χρέος να μείνει σε βιώσιμο επίπεδο ενώ θα ενίσχυε την ικανότητα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Θα γνωρίζετε όμως ότι την Τρίτη το βράδυ το Κυπριακό Κοινοβούλιο απέρριψε αυτό το σχέδιο και δεν δέχτηκε την ε, πρόθεση να υπάρξει επιβολή ενός εφάπαξ φόρου για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο. Η ίδια η πρόταση έδειχνε τις εξαιρετικές καταστάσεις που ισχύουν στην Κύπρο και την ανάγκη να μειωθεί το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τώρα εναπόκειται στις κυπριακές αρχές να υποβάλουν νέες προτάσεις με εναλλακτικέ θέσεις και η Ευρωμάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την Κύπρο στις προσπάθειες μεταρρύθμισης επί τη βάση του συμπεφωνημένου προγράμματος σταθεροποίησης. Πρέπει να είμαι σαφής ότι η Ευρωομάδα ήταν πάντα πεπισμένη και εξακολουθεί να είναι πεπισμένη πρέπει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση των μικροκαταθετών από του μεγάλου καταθέτε και υπογραμμίζει τη σημασία να υπάρξει πλήρη εγγύηση των καταθέσεων κάτω των 100.000 ε, ευρώ. Σας φαίνεται κάπως φιλόδοξο σε μια τέτοια εβδομάδα, αλλά ως νέος πρόεδρος της Ευρωομάδος θέλω να μπορέσουμε στο άμεσο μέλλον να μεταφέρουμε την ατζέντα μας από την αντιμετώπιση των κρίσεων σε μια διαφορετική συζήτηση για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην, στο χώρο του στη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας και ίσως και τις επόμενες φορές που θα συναντηθούμε. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τους βασικούς μας στόχους που είναι η υποστήριξη ισχυρής, βιώσιμης και περιεκτική οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσει απασχόληση και διατηρεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στο οποίο είμαστε όλοι προσιλωμένοι. Πιστεύω ότι όλοι συνενούμε σε αυτά τα εγχειρήματα και του στόχου. Το θέμα είναι πώ θα πρέπει να επιτευχθούν όλα αυτά. Ανησυχούμε όλοι για τι κοινωνικέ συνέπειε αυτή τη κρίση. Είναι μια ενασχόληση που και εγώ συμμεριζόμαι μαζί σα. Όπω είπε η Επιτροπή σα στην έκθεσή τη για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, η κρίση έχει οδηγήσει πάρα πολλούς Ευρωπαίους σε μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε όταν προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις απαντήσεις μας σε επίπεδο πολιτικής. Όπως λέει και η έκθεσή σας, όμως για να μπορέσουμε να έχουμε απασχόληση, ανάπτυξη και να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, θα πρέπει να εξηγιάνουμε τα δημοσία οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι υψηλός λόγος χρέος προς το ΑΕΠ είναι ένα φρένο, μια τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Εμποδίσουν τι επενδύσει οι οποίε μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη, αυξάνουν το κόστο δανεισμού και οδηγούν σε αστάθειε αγορέ. Όπω τόνισε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι και προσιλωμένοι στην εξυγίανση των δημοσιονομικών στι χώρε μα. Αυτό μπορεί να είναι βάρο για την ανάπτυξη σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αλλά είναι προαπαιτούμενο για τη σταθερότητα, η οποία με τη σειρά τη είναι απαράγραπτη για την σταθερή ανάπτυξη στο μέλλον το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και η ε, συνθήκη για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα θα πρέπει να μείνουν ακρογωνία η λύθη της ε, θέσης μας στα δημοσιονομικά. Δίνουν εμπιστοσύνη στους ε, καταναλωτές και στις αγορές και για μένα είναι σημαντικό να γίνουν σεβαστές στην περιοχή του ευρώ. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση των στρατηγικών μόνο επί τη βάση των διαφορετικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρα, αλλά με σεβασμό πάντα των κανόνων του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Τα κράτη-μέλη τα οποία καθυστερούν θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το σύμφωνο. Αυτό απαιτεί να υπάρξει σύντομη διόρθωση των ε, ελλημάτων και βιωσιμότητα σε μακροχρόνιο επίπεδο των δημοσίων οικονομικών. Αυτό κάνουμε και στι κάτω χώρε. Το έλλειμμά μα θα ξεπεράσει τους στόχους εφέτο, γι' αυτό έχουμε εγκρίνει ένα πρόσθετο πακέτο για το έτο 2014, που αφήνει βέβαια περιθώριο για να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας το 2013. Αυτή η Αυτές οι μορφές περικοπής δεν είναι κάτι που στοχεύαμε όλοι μας να κάνουμε ως πολιτική, αλλά στο τωρινό στάδιο είναι αναπόφευκτες και πιστεύω ότι εν καιρό θα αποδώσουν καρπούς. Αν είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη η εξυγίανση των δημοσιονομικών. Παράλληλα όμω πρέπει να κάνουμε διαρθρωτικέ αλλαγέ για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία, τι νέε τεχνολογίε και να αυξήσουμε την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα προσόντα τη εργασιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για του νέου και να του επιτρέψουμε να έχουν πραγματική εμπειρία στον εργασιακό χώρο η κρίση έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέδειξε πόσο αλληλένδετα είναι τα τμήματα της Νομισματικής Ένωσης και πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την ολοκλήρωση <clears throat> της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τόνισα τη σημασία του να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στα δημοσιονομικά και στην οικονομική πολιτική. Αλλά είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Όλα τα θέματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την Τραπεζική Ένωση, φυσικά αυτά είναι στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου Ακοφήν. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Η Συμφωνία για τη Δημιουργία ενό ενιαίου υποπτικού μηχανισμού για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση αυτή. Θα δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στην Ευρωζώνη και τώρα το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι <clears throat> να προχωρήσουμε προς ένα ενιαίο μηχανισμό επίλυσης, ώστε οι τράπεζες οι οποίες δεν ευσταθούν θα μπορούν να επιληθούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι τακτικός και οργανωμένος. Καθώς προχωρούμε σε αυτές τις σημαντικές και μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις στον χώρο του ευρώ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι διαρκεί και συνεχίζεται η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά τη σύγκλωση, σύγκληση των κρατών μελών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ευρώ ως νόμισμά τους. Από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξουν οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τη ε, ζώνη του ευρώ και επομένω να γίνει με σωστό τρόπο η διευνησή του. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονό ότι η Λετωνία ζήτησε να υπάρξει μια έκθεση σύγκληση. Αυτό καταδεικνύει αυτό που γνωρίζαμε ήδη, ότι το ευρώ παραμένει πολύ σημαντικό και πολύ ελκυστικό και βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αυτή είναι κάποια από του τομεί στου οποίου εγώ θα συγκεντρώσω τι προσπάθειέ μου στα επόμενα χρόνια και προσβλέπω στο να ακούσω τι απόψει σα και να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή αρχή. Είμαστε εντό χρονοδιαγράμματο, ε, το οποίο με ικανοποιεί πάντα ιδιαίτερω, ε, γιατί διευκολύνει τη διαχείριση του χρόνου. Α περάσουμε στον πρώτο γύρο ερώτα απαντήσεων. Ζαν Πολ Καουζές, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό και Πρόεδρο του Eurogroup ε, εκ μέρους ε, του ΕΛΚ και μου του Ιδίου. Είπατε ότι υπήρξατε εδώ ε, βοηθός ε, ευρωβουλευτού, όμως σήμερα έρχεστε εδώ με μια διαφορετική ιδιότητα. Δεν θα σας θέσω ερωτήματα ε, ε, για την Κύπρο. Απλώς να πω ότι οι συνθήκες από τις οποίες ε, έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις οδήγησαν στους συμπολίτε μας με εφόσον είχαν αποπροσανατολιστεί και από τον τύπο, να οδηγήσουν ότι πρόκειται για μία διακινδύνευση των καταθέσεων, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για ένα νομισματικό μέτρο φορολογικό μέτρο άλλης φύσης, ε, με φορολόγηση στην πηγή. Τώρα πρέπει να περάσουμε στον ρόλο του Κοινοβουλίου και τη σύνδεσή του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Νομίζω ότι και στη χώρα σας έχετε κάνει δηλώσεις για αυτό το θέμα και θα ήθελα να μάθω τη θέση σας ε, για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ζητήματα που αφορούν το ευρώ, καθώς ε, με αυτό το ζήτημα ασχολείστε κυρίως, και με τον τρόπο ε, διαμόρφωση των συνδέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασιστικό ρόλο να διδραματίσει στο νομοθετικό έργο που αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης, ιδίω ε, σε όλο το έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ΕΚΟΦΗΝ, ε, στην Τραπεζική Ένωση, όλο αυτό το εγχείρημα που απαιτεί ισχυρή δέσμευση και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά αυτό εξαρτάται και από τα εθνικά κοινοβούλια. Οποιουδήποτε είδους ε, συνεργασία ε, μπορεί να υπάρξει μεταξύ των δύο, θα είναι κάτι το ωφέλιμο και θα ενισχύσει την δημοκρατική νομιμότητα των πολιτικών που χαράσουμε στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί ακόμα ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, είτε σε επίπεδο επιτροπών, είτε σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πολ Εντάξει. Ας περάσουμε λοιπόν στο συντονιστή, στην συντονίστρια Ελίσσα Φερέιρα από τους Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Ντέσελμπλουμ που είσαστε μαζί μα. Θα ήθελα να μπορέσω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας αναφέρω και ορισμένε επικρίσεις. Και είναι αναπόφευκτο να αναφερθώ στο θέμα της Κύπρου. Η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι τα 100.000 ευρώ ήταν η μόνη ελπίδα που είχαν οι, Ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι πολίτες ενώπιον της κρίσης. Η απόφαση που ελήφθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σίγουρα έχει υποσκάψει αυτή την εμπιστοσύνη όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω να διαψεύσετε την εντύπωση ότι παρά το γεγονός παρά το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε να υπάρχει ενιαία εποπτεία των ε, ευρωπαϊκών τραπεζών Εξακολουθούν τα κράτη-μέλη να έχουν τη δική τους αντιμετώπιση για τις τράπεζές της και είναι οι καταθέτες οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν την ύφη για να διασώσουν τους μεγάλους πελάτες και τους μεγάλους μετόχους όταν ακόμα και οι τελευταίοι πολλές φορές δεν πληρώνουν καθόλου για τη διάσωση αυτή. <clears throat> Θα ήθελα να ξέρω αν μια ενιαία ε, τραπεζική αρχή και μια ενιαία ε, εποπτική αρχή που ασχολείται και με την επίλυση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ε, φορολογικούς παραδείσους και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρημάτων και αν αυτή θα είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας του Eurogroup. Ευχαριστώ κυρία Φερέιρα για τις ερωτήσεις σας. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτή την εβδομάδα. Άρα είναι πολύ καλό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αμέσως. Αυτό που κάναμε στο Eurogroup μετά από διαδικασία μηνών προετοιμασίας, τις πρώτες συνομιλίες που ξεκίνησαν τον Ιούνιο, θέλαμε να ετοιμάσουμε ένα πακέτο που θα επέτρεπε στην Κύπρο να κάνει μια νέα αρχή, να ακολουθήσει βιώσιμο δρόμο. Τούτου λεχθέντος πρέπει να δείτε ποια είναι η βιωσιμότητα του χρέους, τον επιμερισμό του βάρους, μελλοντική ανάπτυξη και ένα νέο μοντέλο για το τραπεζικό σύστημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Κύπρο. Αυτό βασικά οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είναι κάτι μεγαλύτερο από 10 δις, διότι το συνολικό δάνειο προς την Κύπρο είναι κρισίμου σημασίας για το κατά πόσο θα μπορέσει η Κύπρος να αποπληρώσει το χρέος. Να μπορεί να βρει η Κύπρος ένα νέο οικονομικό μέλλον. Αυτή ήταν το πρώτο βασικό σημείο που ετέθη. Το δεύτερο. Το βιώσιμο χρέος για την Κύπρο σημαίνει χρέος προς ΑΕΠ λόγο όχι παραπάνω από 100. Μετά έπρεπε να έχουμε αναδιαρθρωμένο και υγιή χρηματοστατικό τομέα που θα επέτρεπε μια νέα οικονομική ανάπτυξη για την Κύπρο. Αυτά τα τρία στοιχεία ε, οδήγησαν στο θέμα του επιμερισμού των βαρών. Έπρεπε επίσης να ζητήσουμε δεσμεύσεις και συνεισφορά από την κυπριακή πλευρά περίπου, ύψους περίπου 6 δις. Στην επεξεργασία του πακέτου εξετάσαμε με πολύ προσοχή πού θα ετίθετο το βάρος και θεωρήσαμε δικαιολογημένο το βάρος να το επομιστούν και εκείνοι που είχαν καταθέσεις χωρίς να διαμένουν στην Κύπρο, όχι μόνο αυτοί που διέμεναν στην Κύπρο. Πολλά από τα φορολογικά μέτρα θα επηρέαζαν βασικά τους ντόπιου, ενώ ο τραπεζικός ε, τομέας αποτελείται από πολλούς καταθέτες που δεν διαμένουν στο νησί. Εξετάσαμε λοιπόν και τις μεγάλες καταθέσεις από ανθρώπους που ήταν εκτός Κύπρου, του εξωτερικού. Και το Eurogroup θεώρησε πολύ σημαντικό ότι θα έπρεπε να είναι δίκαιος ο επιμερισμός του, των βαρών και το βάρος που θα επιβάλλεται στι μεγάλε καταθέσει θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που επιβάλλεται στι μικρέ καταθέσει. Εξακολουθούμε να το πιστεύουμε αυτό. Το αποτέλεσμα, η πρόταση, το προτινόμενο πρόγραμμα απερίφθη από το Κοινοβούλιο της Κύπρου. Προσπαθεί η Κύπρος να βρει εναλλακτικέ λύσεις, να καταλήξει στους ίδιους αριθμούς τα ίδια ποσά με διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω πραγματικά να επιτευχθεί μια πιο δίκαιη ισορροπία και αυτό προσπαθήσαμε, σε σχέση με αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε την Παρασκευή το βράδυ. Το Eurogroup πιστεύει ότι πρέπει να είναι δίκαιη η κατανομή των βαρών. Μεγαλύτερη συνεισφορά από τους μεγάλους καταθέτες από ότι από τους μικρότερους καταθέτες. Μετά το σύστημα εγγύησεως καταθέσεων. Αναμφισβήτητα το επιβεβαιώσαμε σαν Υπουργοί Οικονομικών αυτό, ότι το σύστημα εγγύησης των α, καταθέσεων εντός Ευρωζώνης εγγυάται ε, καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Θέλαμε μέσω των, των εισφορών να δημιουργήσουμε βιώσιμο μέλλον για την Κύπρο. Ήταν φορολογικό το μέτρο που προτείνονταν. Ήταν κάτι σαν φόρος εισοδήματος στην αρχή η πρόεδρος έκανε κάποια σχόλια όσον αφορά το πώς παρουσιάστηκε το θέμα, την επικοινωνία. Αναφέρθηκε και στη συζήτηση που κίνησε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί. Βλέποντας τα αυτά έπρεπε από την αρχή να τα έχουμε εξηγήσει περισσότερο. Διάκριση ενός φόρου τέλους από τη μία πλευρά που είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από το να πληγεί το σύστημα εγγύησεως καταθέσεων. Και το σύστημα εγγύησεως καταθέσεων είναι καλυμμένο, θωρακισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών το υπογράμμισαν εκ νέου ε, στην ε, συνέντευξη που δώσαμε τη Δευτέρα, στην ανακοίνωση που κάναμε. Εντάξει, αυτό κάτσε περισσότερο, αλλά είναι βασικό θέμα. Λέει κυρία Μπόλς, πάμε στην Άλντε. Ο Βολφ Κλίτς έχει το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημά μου το εξής. Με ακούτε? Η δική μου κατανόηση είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότερος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακεφαλαιώσει τράπεζες όταν υπάρχει ένας συστημικός κίνδυνος και όταν η επαναπληρωμή των χρημάτων είναι εξασφαλισμένη. Εγώ θα ήθελα να ξέρω κατά τη δική σας άποψη αν θεωρείτε ότι είναι συστημικό το πρόβλημα της Κύπρου, συστημικός ο κίνδυνος. Δεύτερον, ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό ότι η εποπτεία ήταν κάπως χαλαρή και το επιχειρηματικό μοντέλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν είναι βιώσιμο. Χαμηλή φόρη, σχετικά χαμηλή ε, αστυνόμευση και εφαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων. Αυτό είναι γνωστό όχι από τον Ιούνιο του 2012, αλλά και από πάρα πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι το 2011 η Ρωσία έδωσε δάνειο στην Κύπρο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί η Κομισιόν έχει τόσο πολύ καιρό αγνοήσει όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχει δράσει. Τρίτο, το, τα συμφέροντα της ε, Ρωσίας μέσα στο χρηματοοικονομικό σύστημα της ε, Κύπρου να χρησιμοποιήσει την Κύπρο προς τα συμφέροντά της. Πώς βλέπει το Ευρωγκρουπ και η Ευρωζώνη τα θέματα αυτά, τι δυνατότητα η Ρωσία να αναλάβει ένα ενεργό ρόλο για τη χρηματοδότηση των χρεών της Κύπρου. Ε, ε, ε, ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Θα μπορούσα να τα πω στα γερμανικά, αλλά όχι, καλύτερα να συνεχίσω στα, ελληνικά, στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ και επιστρέφω στα αγγλικά λοιπόν τμήμα του προβλήματος στην Κύπρο είναι βεβαίω το τραπεζικό μοντέλο ε, και οι κίνδυνοι με τους οποίους ε, λειτουργούσαν μέχρι τώρα οι τράπεζες και τμήμα της λύσης θα πρέπει να είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και η μείωση του μεγέθου του και η οικοδόμησή του βάσει ενό ε, υγιούς οικονομικού μοντέλου. Είναι αναπόφευκτο αυτό και αυτό είναι τμήμα του προγράμματο και του μνημονίου και των παρατηρήσεων που έχουμε κάνει ε, κατά την εξέταση των ε, ρυθμίσεων για την αποφυγή του ξεπλήματος ε, χρήματος, αν υλοποιούνται όλα αυτά στο πλαίσιο των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν συλλέγονται οι κατάλληλοι φόροι και ούτε καθεξής. Τώρα, γιατί μας πήρε τόσο πολύ χρόνο. Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Εν μέρη, οι φορολογικές πολιτικές παραμένουν εθνική αρμοδιότητα. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν εκεί λοιπόν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί ακόμα να επιληθεί κάτι τέτοιο. Αλλά πράγματι μας πήρε πολύ καιρό. Συμφωνώ μαζί σας. Και οδήγησε σε αρκετού κινδύνους αυτό. Ρωτήσατε αν ε, η Κύπρος αποτελεί συστημικό κίνδυνο. Νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση και με την τρέχουσα όχι αστάθεια, αλλά για τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αστάθεια στην Ευρωζώνη, θα πρέπει πραγματικά να υπερασπιστούμε την ακαιρεότητα της Ευρωζώνης. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση περί συστημικού κινδύνου, αν πρέπει να κάνουμε κάτι από αυτού, αυτομάτως πρέπει να πάμε παραπέρα και να πούμε τι θα κάνουμε για να το επιλύσουμε το πρόβλημα. Έτσι θέλω να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Στην τρέχουσα κατάσταση λοιπόν σίγουρα υπάρχει συστημικός κίνδυνος και η ανησυχία των τελευταίων ημερών αυτό το απέδειξε δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς ένα πρόγραμμα που θα έρει αυτό τον κίνδυνο για την Κύπρο. Μετά, για τον ρόλο της Ρωσίας, όπως ρωτήσατε. Ήδη επισημάνατε ότι υπάρχει ένα δάνειο ύψους 2,5 δις και εν ώψη της ε, συνεδρίασης την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχαν συνεδριάσεις, ε, συναντήσεις και επαφές με τους Ρώσους, τι θα κάνουν ε, για την επέκταση της διάρκειας του δανείου, μείωση του επιτακίου, αλλά <clears throat> για άλλες επιλογές επιπλέον δανείου ή επενδύσεων στις τράπεζες, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τέτοιες κινήσεις. Ε, το μοναδικό που συζητήθηκε στις εβδομάδες πριν από την ε, συνάντηση είναι ότι το δάνειο όσο έχει αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να επιμηκυνθεί. Κατά πόσο θα μπορούσε να επιμηκυνθεί και αν κάτι θα μπορούσε να γίνει για το επιτόκιο. Βεβαίω τώρα η ε, κυπριακή κυβέρνηση έχει συζητήσεις με τη Ρωσία, δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Αυτά εμείς κάναμε κατά την προετοιμασία του πακέτου. Μιλήσαμε με τους ε, Ρώσους για το θέμα του δανείου. Το μόνο που μπορώ να πω πέρα από αυτό είναι ότι αν οι Ρώσοι έλεγαν θα μπορούμε να δανείσουμε κι άλλα, αυτό δεν θα ωφελούσε την βιωσιμότητα του χρέους γιατί η αύξηση του χρέους στην Κύπρο δεν μας βοηθάει να κινηθούμε προς ένα νέο μέλλον. Και αυτό από την αρχή ήταν ο στόχο μας. Δηλαδή να βοηθήσουμε τους Κύπρους να μειώσουν τα προβλήματά τους, ε, να εξηγιάνουν ε, ε, τον χρηματοπιστωτικό τους τομέα και γι' αυτό είπαμε ότι το πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δις. Δάλλος δεν είναι μια βιώσιμη θέση για την Κύπρο, για να κάνει μια νέα αρχή. Ευχαριστώ για τη συντηρητική ομάδα, κύριο Σέπιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω εν, ε, εκ μέρους του ECR και ιδίως... Ε, από την Βελική Αντιπροσωπεία. Ε, ξεκινήσατε πολύ δυναμικά στην Ευρώπη. Πέρσι μας λέγατε βέβαια ότι τα, περισσότερα, τα χειρότερα είχαν περάσει, αλλά μάλλον δεν ισχύει αυτό. Ε, η Κύπρος πλέον είναι η πέμπτη χώρα που έχει λαμβάνει πρόγραμμα διάσωσης και υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και φαίνεται ότι ε, δεν πρέπει να είναι μόνο οι κάποιες χώρες που αναλαμβάνουν το βάρος τέτοιων εγχειρημάτων. Αυτό είναι θετικό. Όμως, βεβαίως το λάθος ήταν η μία απαλλαγή των καταθετών μέχρι τις 100.000 ευρώ. Και αυτό οδήγησε σε διέξοδο. Ε, για μένα το ερώτημα είναι ποιο ζήτησε αυτή τη μία απαλλαγή. Ήσασταν εσείς, ήσασταν ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κύπρος ή όλοι μαζί. Μόλις ε, μιλήσατε για μια ε, δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υπάρχει. Επομένως, θεωρείτε ότι η ισορροπία της Παρασκευής δεν ήταν δίκαιη. Όμως, ε, εσείς ήταν πρόεδρος. Μετά, στην Κύπρο, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα διάσωσης, bailout, γιατί είναι στο τμήμα της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Όμως αυτό δεν ισχύει. Μετά, για την πορεία προς τη Μόσχα ε, ίσως ε, θα πρέπει να μιλήσουμε εδώ για τον κύριο Πούτιν. Ε, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ο, ο γαμπρός μου βέβαια είναι Ρώσος, αλλά να σας πω ότι ο Πούτιν πρώτα θα οδηγήσει την Κύπρο... Ε, θα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη, ας πούμε, και μετά θα... Η Κύπρος θα αποτελέσει ένα είδους σφαίρας επιρροή για τη Ρώσια Ρωσία και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη ε, εκτίθεται και οι Ρώσοι απλά γελάνε. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον κύριο Πούτιν. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Έπινγκ για τις ερωτήσεις σας. Κάνατε σαφές ότι πολλοί από εμά πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει στο τέλος της κρίσης αρκετά πρόσφατα εγώ από την αρχή ήμουν πολύ προσεκτικό να μην κάνω μια τέτοια δήλωση. Είναι αρκετά εύθραυστη η κατάσταση και η τελευταία εβδομάδα έδειξε πόσο πραγματικά εύθραυστη είναι η εμπιστοσύνη που υπάρχει από την πλευρά των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών παρά το γεγονός ότι η ζημιά ήταν περιορισμένη αυτή τη βδομάδα. Αλλά θα ήλπιζα να μπορέσουμε να πούμε ότι έχει τελειώσει η κρίση αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Τονίσατε ότι δεν είναι δικαιωματική η διάσωση. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά υπάρχει και το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον είναι η ενίσχυση της ζώνης του ευρώ, η ενίσχυση του τραπεζικού τομέα σε όλη την ευρωζώνη, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος επιμόλυνσης. Και το κοινό συμφέρον είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, Ευρωζώνη και να την προστατεύσουμε από τη διάδοση της κρίσης. Υπάρχει λοιπόν για αυτό το λόγο μια δέσμευση να βοηθήσουμε την Κύπρο. Είπατε ποιο πρότεινε να υπάρξει ο φόρος για τις καταθέσεις κάτω των 100.000. Εγώ ως πρόεδρος του ε, Eurogroup πρέπει να αναλάβω ευθύνη για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το τάδε θεσμικό όργανο ή το τάδε άτομο. Ήταν μια κοινή απόφαση αν κάποιος πρέπει να πάρει ευθύνη για αυτήν την απόφαση, θα πρέπει να είμαι εγώ. Εγώ υποστηρίζω αυτή την επιβολή φόρου, γιατί είναι ένας τρόπος να ζητήσουμε την ε, συμμετοχή των καταθετών στην Κύπρο, αν ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα πακέτο το οποίο δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπερχρέωση της Κύπρου από τα 10 δισεκατομμύρια που ανέφερα προηγουμένως. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποια επιβολή φόρου στους καταθέτες για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ελπίζω ότι το πακέτο θα είναι ένα δίκαιο πακέτο, όπως και η εταίροι μου στο Eurogroup, θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια κατανομή βαρών με ένα δίκαιο τρόπο. Εδώ αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν. Λέτε αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν σωστή η κατανομή της Παρασκευής. Ήταν δίκαιη με τη μορφή ότι η επιβολή φορολογίας στους μικροκαταθέτες ήταν πιο μικρή από τους μεγαλοκαταθέτες. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει και μεγαλύτερη δικαιοσύνη και μετά από τις ε, επαφές που είχαμε συνεχίσουμε να προσπαθούμε να έχουμε μια προσδοκία λύσης που θα μετακυλήσει περισσότερο το βάρος στους μεγάλους καταθέτες. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχουμε την υποστήριξη και των, ε, της εμπλεκόμενης χώρας και όλων των εμπλεκομένων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι σε κανένα. Είχαμε το αποτέλεσμα της Παρασκευής Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης αμέσως συνέδεσαν αυτό το φόρο με το σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να διαρθώσουμε διαφορετικά το πακέτο και την επιβολή φόρου ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα είναι πιο ισοδικαία. Πάμε στους πράσινους. Άικουτ. Μπες Άικουτ. Ευχαριστώ Σάρων. Καλημέρα κύριε Δέσσερπλουμ, χαίρομαι που είστε εδώ. Κατάλαβα καλά, χθε είπατε ότι προσπαθήσατε να κλείσει το χάσμα μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Βρυξελών και ότι θεωρείτε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ρόλο να ε, κλείσουν αυτό το χάσμα. Βεβαίω, εγώ βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμά μα προβληματίζει το χάσμα εντό ε, τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη μεταξύ των κρατών μελών. Η συζήτηση που υπάρχει στη Γερμανία και στην Κύπρο και το χάσμα μεταξύ των δύο ε, περί αυτού συζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα πρέπει να συζητά και ο πρόεδρος του Eurogroup. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Γερμανία ε, έχει δυσκολίε αυτή τη στιγμή γιατί είναι και έτος εκλογών. Μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά και ε, τα, η μεγαλύτερη συμμετοχή των καταθετών και αυτή μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά ο ρόλο του, του Προέδρου του Eurogroup είναι να συγκεράζει αυτά τα δύο συμφέροντα. Και εκεί ήταν το σφάλμα σας κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να λέτε ότι ε, θα επιθυμούσατε κάτι τέτοιο ή ό,τι θέλετε τέλο πάντων, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι ήταν επιθυμητό οι μικροί καταθέτε να πληρώνουν περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα διάσωση. Ιδίω εσεί ω σοσιαλδημοκράτη, πώ συμφωνήσατε με κάτι τέτοιο. Και ω πρόεδρο του Eurogroup, πώ δεν ε, αντιδράσατε, γιατί δεν αντισταθήκατε. Εσεί είστε υπεύθυνο για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Και αυτή η σταθερότητα δεν υπάρχει υπάρχει στιγμή. Μάλιστα, βάσει των Financial Times, ήταν δική σας η πρόταση ε, να, να πάμε στο 6,70% για τους μικρούς καταθέτες. Ισχύει αυτό. Γιατί δεν αντιδράσατε, γιατί δεν ε, φέρατε αντίρρηση και ποια ήταν τα σφάλματά σας, τι μάθημα αντλήσατε για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Έκχοτ για τις ερωτήσεις σας. Οι παρατηρήσει μου χθε ε, στην Ολλανδία αφορούσε τη δημοκρατική νομιμότητα των όσων εμείς ε, εδώ στις Βρυξέλλες ε, έχουμε κάνει. Να επιστρέψω στα αγγλικά. So, λοιπόν, έκανα κάποιε παρατηρήσει χθε σχόλια όσον αφορά τη συζήτηση τη δημοκρατία στην Ευρώπη, τη δημοκρατική νομιμότητα των όσων εμεί, το Eurogroup, καταρχά, γιατί είμαι πρόεδρο του Eurogroup, αυτών που κάνουμε στην Ευρώπη και εξέφρασα ανησυχίε όσον αφορά αυτό το θέμα και είπα ότι για μένα δεν τίθεται τόσο ζήτημα κατά πόσο πρέπει να συνομιλούν περισσότερο τα κοινοβούλια να επηρεάζουν περισσότερα τα εκτενόμενα. Μεγαλύτερη επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Βεβαίω και αυτό είναι πολύ σημαντικό και χθε είπα ότι θα ήμουν υπέρ μεγαλύτερου ρόλου των κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Το βασικό που είπα είναι ότι δεν φαίνεται να βοηθάει να πετύχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Θεμελιώδες το ζήτημα λοιπόν. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές πολιτικές εν γέννη. Επανακαθορίσατε το ζήτημα εσείς και είπατε ότι είναι θέμα του τι συμβαίνει μεταξύ χωρών. Περισσότερο αυτό μετράει. Εγώ μάλλον διαφωνώ. Γίνεται συζήτηση μεταξύ χωρών και πολλές φορές οι χώρες έχουν πολύ διαφορετικές αφετηρίες και πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Γίνεται και ζωή συζήτηση στην, για την Ευρώπη μεταξύ χωρών. Κοιτάξτε τι, γίνεται, τι έγινε στις Ιταλικές εκλογές. Ήταν βασικό θέμα Ευρώπη. Στις εκλογές στη χώρα μου η Ευρώπη ήταν από τα βασικά θέματα των εκλογών που διεξήχθησαν πέρσι. Ναι, καμιά φορά υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών και τα συμφέροντα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Όμως ε, πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που πετύχαμε ήταν ε, συμβιβασμός όλων αυτών των συμφερόντων. Όπως προανέφερα, ήταν ένα πακέτο που επέτρεπε στην Κύπρο να έχει ένα βιώσιμο χρέος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο το πακέτο, τότε όμως δεν θα βοηθούσε καθόλου την Κύπρο. Ήταν ένας τρόπος να καταλήξουμε σε μικρότερο χρηματοστικό τομέα της Κύπρου, υγιέστερο, χωρίς να καταστραφεί. Υπήρχαν και πιο ριζοσπαστικέ λύσει για την αντιμετώπιση του τομέα. Δεν ακολουθήσαμε το δρόμο. Θέλαμε να ξεκινήσει από την αρχή ε, να κάνει μια νέα αρχή η Κύπρος ε, όσον αφορά το χρηματοδοτικό της τομέα. Αναφερθήκατε στους μικρούς καταθέτες. Είπατε ότι έκανα εγώ λάθος και έπρεπε να σταματήσω αυτή την πρόταση ε, όσον αφορά το να πληρώσουν φόρο οι μικροί καταθέτες. Εγώ επομίζομαι πλήρως την ευθύνη, ήμουν πρόεδρος, είμαι πρόεδρος, αλλά ειδικά τα διάφορα συμφέροντα των διαφόρων χωρών, οι απόψεις και οι θέσεις της ίδιας της Κυπριακής κυβερνήσεως προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία, να μην είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, όλα αυτά οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και σαν Πρόεδρος πρέπει ο Πρόεδρος να συγκεράσει τις απόψεις των διαφόρων χωρών, τις διάφορες οπτικές γωνίες, τους διάφορους κοινού στόχους και γι' αυτό και αν μπορούσα δεν που δεν μπορούσα, δεν, δεν σταμάτησα αυτή την απόφαση, διότι η απόφαση αυτή προσπαθούσε να συγκεράσει όλους τους στόχους και όλα τα συμφέροντα. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Νίκολας, Νίκολας Χουντής. Ένα ερώτημα που δεν απάντησα. Ο κύριος Έικαρτ αναφέρθηκε σε αυτό το άρθρο στο Financial Times ήταν εσφαλμένο, ήταν λάθος αυτό το άρθρο και αυτή η ιστορία. Εγώ σε διαφορετικά ονόματα. Ε, το Financial Times σε διαφορετικές μέρες διάβασα τα διάφορα άρθρα. Ε, λοιπόν, Νίκο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς η πρώτη σας παρουσία συνδέεται με μια απόφαση του Eurogroup που πρώτον αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης και δεύτερο, πράγμα που θα το έχετε αντιληφθεί εσείς και οι άλλοι Υπουργοί Οικονομικών, ότι αυτή η απόφασή σας για την Κύπρο περί φορολόγηση των καταθέσεων έχει δημιουργήσει μια γενικότερη ανασφάλεια στην Ευρώπη, ανασφάλεια των καταθετών, πράγμα που το διαπιστώσατε εδώ. Το λάθος σας τεράστιο. Αναρωτιέται κανείς, εκεί στο Eurogroup είστε ανίκανοι ή έχετε άλλους σκοπούς. Ο κύριος Σόιμπλε δήλωσε ε, σχετικά με τη σχετική απόφαση ότι βεβαίως όποιος επενδύει τα χρήματά του σε χώρες που έχουν λιγότερους φόρους ε, και όπου ελέγχεται λιγότερο όταν οι τράπεζές τους ήταν βιώσιμες θα έχει προβλήματα. Δηλαδή ο κύριος Σόιμπλε ξεκαθάρισε τον ένα στόχο. Φύγετε από τις τράπεζες χωρών αυτών της Κύπρου κτλ. Και, ελάτε στις γερμανικές τράπεζες. Τον άλλον, τον ανομολόγητο στόχο δηλαδή να αγοραστούν δωρεάν το φυσικό αέριο στην Κύπρο όπως και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα δεν το πει. Και τώρα το ερώτημα είναι, επειδή υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο χρηματοπιστωτικός τομέας τους σε σχέση με το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερος από την Κύπρο, πολλοί ρωτούν τι να κάνουν τα χρήματά τους. Ή να σας το πω διαφορετικά, εσείς που καταθέτετε το μισθό σας για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά σας. Και το ερώτημα που υπάρχει είναι υπάρχουν χώρε όπου κινδυνεύουν οι καταθέσεις των αποταμιευτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Χούντι. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το σύστημα εγγύησεως των καταθέσεων και η εγγύηση μέχρι 100.000 είναι απόλυτη και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει πρόθεση να φυγεί. Αυτή είναι μια συμφωνία που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν οποιαδήποτε χώρα σε οποιαδήποτε περίπτωση ε, θέλει να θέσει το σύστημα αυτό εφαρμογή, σε εφαρμογή των, ε, της εγγύησης των καταθέσεων είναι ευθύνη της χώρας που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα να αποζημιώσει τους καταθέτες. Τώρα μια εφάπαξ εισφορά για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των τραπεζών όπως στην περίπτωση της Κύπρου αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδύρυτο, είναι αναπόφευκτο άμα δείτε την κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου και αν συμφωνήσετε ότι ένα πακέτο που θα ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια, ένα πακέτο διάσωσης, δεν θα έδινε καμία δυνατότητα ανάκαμψης στην Κύπρο. Στην προσπάθεια λοιπόν εξισορρόψης ενός πακέτου το οποίο θα επέτρεπε να υπάρξει ένα νέο μέλος στην Κύπρο και συγχρόνως να υπάρξει μια συνεισφορά από την ίδια την κυπριακή οικονομία ήταν αναπόφευκτο, τουλάχιστον κατά την άποψη του Eurogroup, ότι θα υπήρχε κάποια συμβολή των καταθετών. Αυτό νομίζω ότι είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω στο ερώτημά σας. Και το αν είμαστε ανίκανοι ή όχι, αυτό θα το αφήσω σε εσά να το κρίνετε. Εντάξει, λέει η πρόεδρος. Ξαναγυρίζουμε στο ΕΛΚ και την κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ναι, Κυρία Πρόεδρε, επειδή είμαι ο μόνος μη εγγεγραμμένος, μήπως μπορώ να έχω το λόγο εξ ονόματος του μη εγγεγραμμένου. Βεβαίω, δεν το είχατε αναφέρει ότι θέλατε να λάβετε το λόγο. Υπάρχει μια διαδικασία. Λυπάμαι πολύ. Νόμιζα ότι ανοίγατε, αφήν, τη συζήτηση για τις πολιτικές ομάδες, επομένως θα είχα τη δυνατότητα να λάβω το λόγο. Εντάξει, λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Καλημέρα κύριε Ντέσερπλουμ. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ με την ε, αποφασιστικότητά σας, γιατί βλέπω ότι είχατε δύσκολες εβδομάδες τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά τις ε, αποφάσεις του Eurogroup τώρα. Τι, πώς θεωρείτε ότι κατεμερίστηκε και πώς ήταν ε, ε, η χρονική στιγμή που ελήφθη αυτή η απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη ε, των καταθετών και κατά πόσο αυτή η εισφορά έθετε σε κίνδυνο την εγγύηση των καταθέσεων. Είπατε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ότι δεν θα μπορούσατε να αποφύγετε κάτι τέτοιο. Ε, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευθεί σε άλλες χώρες. και έθεσε και ένα ερώτημα εδώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τώρα, να περάσω στο εξή. Η Κύπρος φαίνεται ότι ανακοίνωσε ότι ε, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κρατικοποίηση των συνταξιδοτικών ταμείων. Αυτό είναι ιδιαίτερα δραματικό γιατί σε ορισμένες ε, χώρες ε, κάποιοι δεν έχουν καν πρόσβαση στη σύνταξη, ε, όπως στις κάτω χώρες. Ε, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Τρίτο ερώτημα. Η Κεντρική Τράπεζα της ε, Κύπρου έχει σταματήσει τη τραπεζική δραστηριότητα στην χώρα, ενώ δεν υπάρχει καμία πτώχευση τραπέζας, τουλάχιστον επισήμως για να αποφευθεί η ανάληψη κεφαλαίου και μεταφορά κεφαλαίων. Ποια είναι η δική σας ε, θέση ως προς αυτή την ε, ε, παράβαση. Μετά, όπως αναφέρθηκε, ότι είναι σφάλμα αυτή η κίνηση κατά της μεταφοράς των εσωτερικών κεφαλαίων και μου φαίνεται και μία έκκληση προς τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Πώς το αξιολογείτε αυτό. Υπάρχει μια φήμη ότι ήδη πολλά κεφάλαια έχουν αποδημήσει από την ε, Κύπρο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και ποια είναι η δική σας άποψη. Και τελευταίο ερώτημα. Είπατε ότι ο Κύπρος δεν πρέπει να λάβει πάνω από 10 δις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τα επιστρέψει. Στην Ελλάδα το δάνειο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Επομένως θεωρείτε ότι ήταν λάθος στην Ελλάδα. Και Τέλος, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ε, για την ε, φορολόγηση, επιβεβαιώνεται ότι αυτό θα ε, συμπεριλαμβάνει και μία αλλαγή του ποσού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρατε σχεδόν όλο το χρόνο, αλλά δεν θα πάρετε απαραίτητα και απαντήσεις, όλες τις απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας, ενώ τρέχει ο χρόνος. Το πρώτο ερώτημά σας. Ευχαριστώ για την ανησυχία σας. Με ρωτήσατε πόση πίεση ε, δέχτηκα όσον αφορά το πρόγραμμά μου. Βέβαια, μεγάλη πίεση επί του παρόντος. Θα καταφέρω μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Δεύτερον, λάθος αναφέρατε αυτά που είπα αυτά που υποτίθεται ότι είπα στο Εθνικό Κοινοβούλιο σαν Υπουργό Οικονομικών, όπου μίλησα χτε για την Κύπρο σαν Υπουργό Οικονομικών. Με ρώτησαν οι σοσιαλιστές στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Ερώτηση λοιπόν. Πώς να το πω. Σκέφτομαι τώρα την Ολλανδική συζήτηση και πρέπει να μεταφράσω στο μυαλό μου τα, από τα Ολλανδικά. Λοιπόν, το έκανα ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα δεν είχε καμία σχέση με το σύστημα εγγυήσεω καταθέσεων. Βέβαια, δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση, το καταλαβαίνω. Δεύτερον, ότι η κατάσταση στην Κύπρο είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Πάρα πολύ προβληματική όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα κλπ. Οπότε, όχι, δεν θα υπήρχε παρόμοιο πακέτο και παρόμοια προσέγγιση για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ήμουν πολύ ξεκάθαρο όσον αφορά αυτό το θέμα. Ρωτήσατε κατά πόσο η, τα μέτρα που ελήφθησαν, όπου κλείσαν οι τράπεζες, ότι επιτρέπεται, έχει όριο ανάληψης κάθε μέρα για κάθε καταθέτη από τα αυτόματα μηχανήματα. Κατά πόσο, όπως το λέμε, είναι, αποτελεί αυτό παραβίαση της ελεύθερης μετακίνησης, διακίνησης ε, κεφαλαίων. Ξαφνικά αρχίζω και χάνω τα αγγλικά μου. Όχι, δεν νομίζω ότι αληθεύει είναι εντό όλων των διαθεσίμων ε, νομικών πλαισίων. Μπορούμε να δράσουμε όταν υπάρξει τραπεζική κρίση. Είναι εν μέρη εθνικό μέτρο και εν μέρη ευρωπαϊκό. Η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα, η Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα έχει νομικά μέσα να κλείσει τις τράπεζες αν υπάρχει κατάσταση ανησυχίας και πανικού στον τραπεζικό τομέα και αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για να ε, ηρεμήσει η κατάσταση και για την ώρα στην Κύπρο γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί ένας τρόπος να ανοίξουν σταδιακά οι τράπεζες ξανά ενώ όσο γίνεται πιο γρήγορα θα κινηθούμε προς ένα τελικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ διότι περάσαμε κατά ένα λεπτό το διαθέσιμο χρόνο. Κόριν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μας εκπλήσει η κυρία Ντάσερ Μπλουμ ε, που ορισμένοι συνάδελφοι προσπαθούν να κάνουν ε, αυτή τη συζήτηση, μια Ολλανδική συζήτηση. Εδώ βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, βεβαίως ε, ε, δεν είναι εύκολη η αρχή σας, πρέπει να ακολουθήσετε στα βήματα του Ζαν Πολ Γιούνκερ και οι πρώτες σας μέρες ήδη έχουν χαρακτηριστεί από ένα αποτυχημένο πρόγραμμα διάσωσης. Όμως ε, είστε και πολύ έμπειρος πολιτικός και βουλευτής Επομένω, ε, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρετε να βρείτε μια καλή λύση. Και για μένα μια καλή λύση δεν είναι, μια μη ρωσική, μια ευρωπαϊκή λύση με ευρωπαϊκές ε, προϋποθέσεις. Και πρέπει να σας επενέσω που εσείς λάβατε την, αναλάβατε την ευθύνη ε, για την αποτυχία του προγράμματος διάσωσης. Γιατί μέχρι τώρα έχω μόνο ακούσει συναδέλφους σας που λέγανε ότι όχι, εγώ δεν είμαι υπεύθυνο. Ακόμα και οι Υπουργοί Οικονομικών ε, που ε, υπερψήφισαν την πρόταση ε, στο Eurogroup δεν ανέλαβαν την ευθύνη που τους αναλογεί. Επομένω, πρέπει να σας συγχαρούμε γι' αυτό, να σας επενέσουμε και να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα ακόμα για αυτούς τους μικρούς καταθέτες ίσως από νομικής πλευράς έχετε δίκιο ότι δεν ε, επλήγει το ε, σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Όμως οι πολίτες δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Και στο μέλλον, αν είναι απαραίτητο, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, ε, τότε πώς ακριβώς θα επιληθεί το πρόβλημα. Γιατί εγώ πραγματικά είναι κάτι με απασχολεί, ότι οι κίνδυνοι για τις τράπεζες είναι μετά ακόμα μεγαλύτεροι. Ε, υπάρχει ο νόμος ε, παρέμβασης, ευρωπαϊκής παρέμβασης ε, και αυτό κατά τη γνώμη μου συμβαίνει ότι οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και οι καταθέτες πρέπει να είναι απολύτως ε, ασφαλείς. Και πώς θα το προσεγγίσετε σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, την εποπτεία των ε, τραπεζών που συμφωνήσαμε την, επί το οποίο συμφωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτω ώστε να υπάρχει άμεση στήριξη από το Ταμείο. Θα ήθελα λοιπόν τις δικέ σα απόψεις από αυτόν. thank you. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Μιλήσατε για ένα αποτυχημένο πακέτο Βλέποντας την κατάσταση αυτή, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν έγινε δεκτό το πακέτο αυτό και οι κυπριακές αρχές αναζητούν ένα εναλλακτικό πακέτο. Εάν αυτό είναι δυνατό μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει και το αν αυτό θα το κάνει βιώσιμο, αυτό δεν έχει νόημα να το ρωτάτε. Εμείς είπαμε ότι θα δώσουμε χρόνο στους Κυπρίους να προτείνουν νέες Κατευθύνσει, αλλά θα πρέπει να είναι υγιεί από οικονομική άποψη και βιώσιμε και φυσικά πολιτικά εφικτέ αυτέ οι προτάσει. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το πακέτο που αποφασίστηκε την προηγούμενη, προηγούμενη Σαββατοκύριακο έχει αποτύχει γιατί δεν υπάρχουν πολλέ δυνατότητε. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εισφορά και είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικέ παραλλαγέ για τη διάρθρωση αυτών των εισφορών από του καταθέτε. Μιλήσατε για τους κινδύνους μιας συρροής καταθετών να αποσύρουν τα χρήματά τους και για το γενικό πρόβλημα πώς αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες που είναι σε δυσκολίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Κοφίν. Αποφασίσαμε να υπάρξει ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Ναι, ναι, έχει τελειώσει αυτό. Σας ευχαριστώ και για την συμμετοχή σας στα θέματα αυτά. υπήρξε μια συμφωνία ότι μέσα στον επόμενο χρόνο μπορεί να γίνει η εκκίνηση του εποπτικού έργου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μηχανισμό επίλυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε ισχυρά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις τράπεζες οι οποίες έχουν προβλήματα. Και έχετε δίκιο, ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή των μετόχων και των ομολογιούχων σε αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα. Αν μπορώ να μιλήσω σαν Ολλανδός υπουργό Οικονομικών, χρειάστηκε να εθνικοποιήσουμε μια τράπεζα στις κάτω χώρες και ήταν ατυχές για τους ε, μετόχους, αλλά έπρεπε ουσιαστικά να εκμηδενήσουμε το μετοχικό του κεφάλαιο είναι ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εργαλειοθήκη. Συμφωνώ ότι πρέπει να επεξεργαστούμε αυτά τα εργαλεία και να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Για την άμεση επανακεφαλαιοποίηση στην Ευρωομάδα, εξετάζουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει να γίνει αυτό πραγματικότητα. Πριν από το καλοκαίρι ελπίζουμε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η άμεση επανακεφαλαιοποίηση για το ΕΛΚ, ο Γκίναρ Χόκμαρκ, ο οποίος είναι και ο εισηγητής για την οδηγία ανάκτησης και αυτή έχει φυσικά κάποια επίπτωση στα, στα πρόσφατα γεγονότα. Ναι, κατανοώ ότι είχαμε πολλή συζήτηση για το θέμα της Κύπρου σήμερα και μπορώ μονάχα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση και όχι μια ρωσική λύση στο πρόβλημα της Κύπρου, αλλά η οποία θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη και στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Βρισκόμαστε πιστεύω στο στάδιο αυτό όταν πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη που αναφέρατε. Και θέλω τώρα να σταθώ σε ένα άλλο τμήμα της παρουσίασής σας κύριε Πρόεδρε. Εσείς τονίσατε την ανάγκη να υπάρξουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι μυστικό το ότι δεν είσαστε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ ότι μιλάμε και λέμε πάρα πολλά αλλά δεν κάνουμε τίποτα για όλα αυτά τα προβλήματα. Ένας από τους λόγους που δεν κάνουμε τίποτα είναι ότι δεν τηρούμε τους πραγματικούς κανόνες που έχουμε. Δεν μιλάμε για το σύμφωνο σταθερότητα. Το σύμφωνο σταθερότητα, εάν υποσκαφθεί, αν υπονομευθεί και χαθεί η αξιοπιστία του, θα έχουμε χρηματοπιστωτικά και δημοσιονομικά προβλήματα και έλλειψη μεταρρυθμίσεων. Επομένως, δεν θέλω να σας μιλήσω μονάχα για την Κύπρο, αλλά για μια πιο μεγάλη χώρα στην Ευρώπη που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου δεν εφαρμόζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και αναβάλει την εφαρμογή των κανόνων για το έλλειμμα. Τι θα κάνετε εκεί. Αν δεν δράσετε, υπονομεύετε και πάλι την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτό το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας για να υπάρξει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, αλλά επίσης και για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο έδαφος και την κατάλληλη ορμή για μεταρρυθμίσεις. Αν εμείς εξακολουθήσουμε να αναβάλουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αναβάλουμε και την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση και οι κοινωνικές συνθήκες που αναφέρατε θα είναι ακόμα οξύτερες. Είσαστε σε μια κεντρική θέση για τα θέματα αυτά. Ακούσατε τις απόψεις και τις επικρίσεις για την πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup. Και εδώ όταν πρόκειται για μια πιο μεγάλη οικονομία, διακυβεύονται πολύ περισσότερα αν υπάρξει λανθασμένη αντιμετώπιση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσετε προβλήματα σε χώρες πολύ μεγαλύτερες από την Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Χέρκμαρκ για το ερώτημα αυτό, για τα ερωτήματά σας καλύτερα και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο άτομό μου όταν μιλάτε για τα μεγάλα προβλήματα στις μεγάλες χώρες. είναι απαραίτητο για μένα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη, να κάνουμε κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και καταλαβαίνω την αδειμονία σας. Από την άλλη μεριά όμως, η κρίση μας έχει οδηγήσει σε κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάποιες χώρες, ακόμα και στη δική μου χώρα, μεταρρυθμίσεις που χρόνιζαν, που είχαν Μα δεν αναφερόμουν στη δικιά σας χώρα, λέει ο κ. Χέκμαρ. <clears throat> Όχι, αλλά είναι πιο εύκολο για μένα να πάρω το παράδειγμα της δικής μου χώρας. Πολλές μεταρρυθμίσεις διαφορετικού χαρακτήρα είχαν καθυστερήσει πολύ στις κάτω χώρες και το οικονομικό μας πρόβλημα τώρα έχει να κάνει με τη στεγαστική αγορά, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πριν από 10-20 χρόνια. Αυτό είναι μια ειλικρινής απάντηση και αυτό αφορά πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχεδόν όλες τις χώρες και εδώ δεν είναι θέμα βορρά εναντίον νότου και γι' αυτό αναφέρομαι στη δική μου χώρα. Έχουμε πραγματικά διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε καθυστερήσει την αντιμετώπιση του για πάρα πολύ καιρό. Η κρίση τώρα έχει ασκήσει πίεση και έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική όθηση να υπάρξει κάτι. Η κρίση τώρα φαίνεται ότι μειώνεται και ελπίζουμε ότι αυτό είναι πραγματικότητα και επομένως μειώνεται και η πίεση για μεταρρυθμίσεις. Δημιουργήσαμε πολλούς νέους μηχανισμούς, που δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί. Μηχανισμοί βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη σε διακυβερνητικό επίπεδο θα πρέπει να έχουν επαφές μεταξύ τους και να λένε το ένα στο άλλο δεν αντιμετωπίζετε την αγορά εργασία σας, δεν βελτιώνετε την ανταγωνιστικότητά σας και αυτό αφορά και το δικό μου χώρο. Αυτό δημιουργεί κινδύνους και για μένα. Επομένως, το να έχουμε μια θέση από κοινού των θεμάτων αυτών, να συζητούμε για την αγορά εργασία, για την οικονομική μεγέθυνση σε κάθε χώρα, να μπορούμε να μαθαίνουμε ένα από τον άλλο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά συνδέονται και με το Σύμφωνο Σταθερότητα. Αν χώρε όπω οι κάτω χώρε, θα μου επιτρέψετε να μιλάω για αυτή τη χώρα, και όχι την άλλη που είναι πιο κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αν χώρε όπω οι κάτω χώρε δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο του κάτω από τα ελλείμματος. Τότε θα πρέπει να έχουν πολύ καλή επιχειρηματολογία για να εξηγήσουν γιατί δεν μπορούν να τηρήσουν τους στόχους και βρισκόνται σε επίπεδο υπερβολικού ελλείμματος. Θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες στην οικονομία τους και θα πρέπει να είναι έτοιμες να καταδείξουν ότι θα προχωρήσουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να πετύχουν στα επόμενα 2-3 χρόνια τους στόχους αυτούς. Ότι θα κάνουν διαφορετικές αλλαγές για να πετύχουν να βελτιώσουν την κατάσταση και σε αυτές τις εξαιρετικές οικονομικές περιστάσεις χρειάζονται έκτακτα μέτρα για να μπορέσει κανείς να επανέλθει στο σωστό δρόμο και μια πιστική επιχειρηματολογία ότι μπορούν να επιτευχθούν αυτά. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε για ορισμένε χώρε ένα πρόσθετο χρόνο για να πετύχουν του στόχου αυτού. Αλλά αυτή η δοκιμασία πρέπει να είναι μεμονωμένη και αυστηρή. Τι θα κάνετε λοιπόν με τη Γαλλία, λέει ο κ. η Γαλλία όπως και οποιαδήποτε άλλη χώρα θα αντιμετωπιστεί επί τη βάση αυτών των κριτηρίων. Αν μπορούν να πετύχουν τους τεθειμένους στόχους σε δημοσιονομικό επίπεδο εφέτος, αν όχι τι μπορούν να κάνουν για να πετύχουν τους στόχους αυτούς το ταχύτερο να για τον, τον επόμενο χρόνο, τι θα κάνουν σε επίπεδο διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων και αυτό ισχύει για τη Γαλλία όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη σύνοψη του Six Pack. Λοιπόν, πάμε στο S&D και τον Peter Σίμον που είναι εισηγητής για το σύστημα εγγύησεως των καταθέσεων και της σχετικής ε, προτάσεις για το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντέσελμπρουμ, θέλουμε αλήθεια και διαφάνεια είναι απαραίτητο να ξέρει ο καταναλωτής όχι τι λέει η συσκευασία, αλλά τι είναι το εσωτερικό της πρότασης. Εγώ θα ήθελα να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα οποία λέτε. Λέτε ότι το πακετάρισμα είναι τέτοιο που να μιλάμε για μια έκτακτη φορολογία. Μπορεί οι δικηγόροι και οι νομομαθείς να το πιστέψουν. Τι πιστεύει όμως ο κόσμος, τι καταλαβαίνει ο κόσμος όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Λένε όχι, δεν μας ενδιαφέρει το περιτύλιγμα, μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι ότι είπατε ότι αν χρεοκοπήσει μια τράπεζα μέχρι 100.000 ευρώ θα πάρουμε πλήρη αποζημίωση. Και τι κάνετε εσείς, το αφαιρείτε αυτό. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ποια είναι η επιχειρηματολογία σας. Όλοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη θα μάθουν ότι οι υποσχέσεις σας αυτές δεν είναι αξιόπιστες. Αλλά η εμπιστοσύνη όπως ξέρουμε είναι το πιο σημαντικό αγαθό. Ο κύριος Γιούγκερ ήταν εδώ παρόντες, παρόν στο παρελθόν και ξέρει ότι ο κύριος ε, Σόιμπλε είχε πει τα ίδια πράγματα που λέτε εσείς. Λέτε ότι είναι μια μοναδική περίπτωση, ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Μην κάνετε το ίδιο σφάλμα. Το ίδιο είχατε πει και για την Ελλάδα. Δεν σας πίστεψε κανένας και τώρα δεν σας πιστεύει κανένας. Δεν πίστεψε το Eurogroup ό,τι και να κάνετε μόνο όταν ο Ντράγκη είπε ότι θα έχουμε απεριόριστη παροχή ρευστότητα, τότε το πίστεψαν οι επενδυτέ. Αν εσεί υπονομεύσετε την εμπιστοσύνη των καταθετών, δεν θα υπάρξει κανένας Μάριο Ντράγκη ο οποίο να μπορέσει να το ανατρέψει αυτό. Εσείς ως Ντάισελμπλουμ είσαστε υπεύθυνο γι' αυτό και όχι οι Κύπροι για το γεγονός ότι δεν πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτή η εμπιστοσύνη. Εσεί θα ήσασταν υπεύθυνο, να πείτε φίλοι στου Κύπριους δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να δίνετε την εντύπωση ότι η Κύπρο μόνη τη μπορεί να αποφασίσει. Γιατί τότε βρίσκεστε εσεί, γιατί βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκεί και ενώ στην περίπτωση τη Ελλάδο ή της Πορτογαλίας τους επέβαλαν θα κάνετε αυτό, εκείνο και εκείνο. Λοιπόν, εσεί πρέπει να ξέρετε τι είναι σωστό και τι είναι λάθο. Εσεί μιλάτε ότι υπάρχει περιθώριο επιλογής το οποίο θα θέσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο. Σε κανένα άλλο δεν δώσατε τέτοιο τράτο για να αποφασίσει. Και δεν μπορείτε να πείτε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση μπορεί να σώσει τους μεγάλους καταθέτες. Όταν υπάρχουν τόσα ε, δισεκατομμύρια στην Κύπρο, έχουν πάρει οι μεγαλοκαταθέτες αν είχε κανείς ένα ένα εκατομμύριο θα είχε πάρει μέσα στα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερους τόκους από ό,τι θα είχε πάρει αν τα είχε βάλει στην Γερμανία. Γιατί λοιπόν δεν τα παίρνετε τα λεφτά από τους μεγαλοκαταθέτες και τα παίρνετε από τους μικροκαταθέτες στην Ευρώπη. Ε, ε, Σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Έχω πλήρη επίγνωση. Ξέρω πολύ το ότι εγώ σε αυτή τη θέση σαν πρόεδρος του Eurogroup πρέπει συνεχώς να δουλεύω στον τομέα της εμπιστοσύνης του κόσμου και ο μόνος τρόπος που αν το πετύχουμε σαν ε, πολιτική είναι να λέμε την αλήθεια και να υπάρχει, να δημιουργούμε σαφήνεια. Αυτά ήταν και αυτά που αναφέρατε, οι δύο βασικές λέξεις που χρησιμοποίησατε και συμφωνώ απόλυτα. Αλήθεια, σαφήνεια. Άρα, η Κύπρος Χρειάζεται ένα πρόγραμμα από την Ευρωζώνη για να βγει από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να δώσει αυτή την υποστήριξη, αλλά για να είναι βιώσιμη η λύση χρειάζεται ένα στοιχείο επιμερισμού των βαρών πλευρά Κύπρου. Το θέμα είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Πώς μπορεί να επιτευχθεί με έναν τρόπο που να μπορεί να το αντέξει ο κυπριακός λαός να είναι δίκαιη η μέθοδος. Και όλοι συμφωνούμε ότι δίκαιο σημαίνει ότι οι μεγάλες καταθέσεις συμμετέχουν πολύ περισσότερο σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι μικρές καταθέσεις. Εξετάσαμε πολλών ειδών φόρους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το πακέτο και το πρόγραμμα. Πολλοί από τους φόρους που εξετάσαμε και κάποιοι αυξάνονται στο πρόγραμμα όπως γνωρίζετε κυρίως ε, πλήττουν τους ντόπιου. Και θεωρήσαμε ότι ήταν δίκιο και ελπίζω να συμφωνείτε ότι θα έπρεπε ε, να ζητήσουμε επίσης δίκαιο, ε, δίκαια συμμετοχή και από τους καταθέτες που δεν διαμένουν στην Κύπρο και συζητήθηκε πώς θα πρέπει, από τι πρέπει να αποτελείται ο φόρος και καταλαβαίνω τις επικρίσεις που εκφράστηκαν όσον αφορά το θέμα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα, είτε της Παρασκευής το πρωί, είτε χρειαζόμαστε και ένα μήνα παραπάνω και δύο μήνες παραπάνω, οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα έπρεπε να το υποστηρίξουν όλα τα κράτη-μέλη και η ίδια η Κύπρος και όταν λέτε μη δίνετε στον κόσμο περιθώρια λιγμών, φοβάμαι ότι δεν πάει έτσι το πράγμα, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στο Eurogroup. Πρέπει να δίνουμε στον κόσμο χώρο, περιθώριο λιγμών. Αλλά ναι, είναι πρόθεσή μα να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατό στη συμφωνία και ναι, προσπαθούμε να βρούμε τρόπου για να ε, καταλήξουμε σε πιο δίκαιη λύση. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα ε, στο ΕΛΚ. Ε, κύριο Θαλμπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωγκρουπ. Νομίζω πέρασαν οι πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης και θέλω να εξάρω τις θυσίε και τις προσπάθειες που έκαναν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από το θέμα της Κύπρου, όπου τα πράγματα μπορούσαν να τα καλύτερα, εγώ έχω εμπιστοσύνη Πιστεύω ότι πρόκειται μονάχα για μια καλοκαιρινή θύελα και όχι για ένα πραγματικό θέμα. Έχουμε τα εργαλεία αυτά όπως και η δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας να δίνει απεριόριστη ρευστότητα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη ε, όλων των εμπλεκομένων και να μην τεθεί αυτό ένα αμφιβόλο. Για μας η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Μιλάτε για μεταρρυθμίσεις. Κάποιες χώρες έχουν καθυστερήσει, άλλες χώρες έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι μονάχα ένας πυλώνας της ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ο άλλος πυλώνας είναι η Ευρωμάδα. Τι θα κάνει η Ευρωμάδα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μια ισορροπία η οποία θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μας, αλλά συγχρόνως και τα απαραίτητα κίνητρα για τη δημιουργία θέσεως απασχόλησης. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά την Τραπεζική Ένωση. Είπατε σε δύο περιπτώσεις ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο πυλώνα στην Τραπεζική Ένωση, δηλαδή τον ενίο μηχανισμό επιλύσεων. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας αλλά η κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι μια ευκαιρία για να δώσουμε πραγματικά μια όθηση προς την κατεύθυνση αυτή, να προχωρήσουμε για να θέσουμε τις βάσεις αυτού του τρίτου πυλώνα της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, του Κοινού Ταμείου ε, Προστασίας των Καταθέσεων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι εκεί φτάνουν τα σπανικά μου. Muchas gracias. Πολύ σωστά είπατε ότι τώρα έχουμε πολύ περισσότερα εργαλεία από ό,τι στην αρχή της κρίσης. Και υπάρχει μια παλιά ρίση που λέει ποτέ μην αφήνεις μια κρίση να πάει χαμένη και νομίζω ότι δεν το κάναμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει πολύ περισσότερα μέσα, μηχανισμούς ε, στη διάθεσή της για να αντιμετωπίζει προβλήματα και συμμερίζομαι και εγώ την ελπίδα σας ότι η τρέχουσα κρίση που αφορά την Κύπρο θα επιληθεί σύντομα. Το κύριο ερώτημά σας ήταν ποια είναι η στρατηγική για την ε, ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι βασικό ζήτημα να αντιμετωπίσουμε την ε, ευαισθησία των των ε, οικονομιών μας. Και έχετε δίκιο ότι σε πολλές ε, χώρες έχουν καταβληθεί πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η Ισπανία είναι μία από αυτές τις χώρες, αλλά και η Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία. Πολλά έχουν γίνει. Και βεβαίως ήταν πολύ μεγάλο το κοινωνικό κόστος, πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό και να είμαστε ειλικρινεί, είμαι σίγουρο ότι η ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών έχει ενισχυθεί και αυξάνεται καθημερινά. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη και τι νέε θέσει εργασία. Δεύτερον, πρέπει συνολικά όλοι μαζί να εργαστούμε για να βρούμε έναν καλύτερο, πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο για την εκτέλεση των προπολογισμών μας. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε νέα μέσα, νέες γραμμές προπολογισμού για την καινοτομία, την εκπαίδευση, ε, ε, την καλύτερη παιδεία για τους ε, νέους, να έχουν καλύτερα πτυχία, να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω μαθητιών και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα σημεία και έχω και επίγνωση του γεγονότος ότι το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα έκανε την απασχόληση των νέων βασική προτεραιότητα και υπάρχει δέσμευση να, να γίνουν επενδύσεις ακριβώς στους νέους και στην απασχόληση των νέων. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην Τραπεζική Ένωση και στον Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών. αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για, αν χρειαζόμασταν μάλλον κίνητρα για να εργαστούμε περισσότερο και πιο εντατικά, η Κύπρος σίγουρα ήταν ένα τέτοιο κίνητρο. Όμως, για να υπάρξει μια τέτοια βιώσιμη αηφόρο οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια τραπεζική ένωση. Είμαι απόλυτα πεπισμένο γι' αυτό. Ένα από του μεγαλύτερου κινδύνου αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχυθούν και οι ισολογισμοί τους, η υποπτία θα πρέπει να ενισχυθεί βεβαίως. Τέτοιοι μηχανισμοί ε, εξυγίανσης θα πρέπει να συσταθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, των προβληματικών τραπεζών. Χρειαζόμαστε εργαλεία ανακεφαλοποίησης και τέλος πρέπει να εξετάσουμε και το σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ήδη πολλοί θεωρούν ότι είναι ευρωπαϊκό μηχανισμό. Όμω το μόνο το οποίο έχει θεσπιστεί είναι αυτό για τι 100.000. Όμω και πάλι είναι εθνική αρμοδιότητα. Ε, να μπουν τα χρήματα εκ των προτένων στο τραπέζι όταν υπάρχει ε, πρόβλημα με τις τράπεζες και ε, στην τρέχουσα κατάσταση ήδη είναι ακόμα μάλλον ένα πολύ, μεγάλο, πολύ ευάλωτο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά, να το υπερασπιστούμε γιατί είναι απόλυτα θεμελιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, ε, στις Τράπεζε και στο τραπεζικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους σοσιαλιστέ. Λία Μουαγκόκ. Καλημέρα Πρόεδρε, καθώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνεται μια συζητή, συζήτηση ηθελογικού τύπου όσον αφορά της Κύπρου, το θέμα της Κύπρου κατά πόσο υπονομεύεται το σύστημα εγγύσεως των καταθέσεων, κατά πόσο γίνεται κάποιο φορολόγηση στην πηγή των περιουσιακών στοιχείων και κάποια, κατά πόσο υπονομεύεται η ελεύθερη μετακίνηση, διακίνηση κεφαλαίων. Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψή του, ζητήθηκε η άποψή του, αρμόδιος Επίτροπος. Από τι πληροφορίε ε, που έχω, μόνο το βράδυ Σάββατο προς Κυριακή ενημερώθηκε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερο ερώτημα αυτό το επεισόδιο δημιουργεί ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα διακυβέρνησης, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα διακυβέρνηση Ευρωζώνης. Το μνημόνιο που για την Κύπρο εμπεριέχει και άλλες προτάσεις όπως ιδιωτικοποίησης και σχετίζεται με αυτό που αρχίζουμε να αποκαλούμε στην Ευρώπη μακροαιρεσιμότητα. Και χθε δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχετικό έγγραφο η μακροαιρετη... αυτή η αν εφαρμοστεί και είναι κάποιοι που την επερασπίζονται στο Συμβούλιο από ό,τι κατάλαβα θα δημιουργεί ένα πρόβλημα νομιμότητας δημοκρατικής έναντι των συμπολιτών μας που είναι πολύ... Ε, έχω μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά τις συστάσεις που κάνει το Συμβούλιο σήμερα. Ποια είναι η άποψή σας. Θεωρείτε ότι αυτή η μακροαιρεσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης διακυβερνητικής ή θέλετε να χρησιμοποιούνται περισσότερο κοινοτικέ μέθοδοι, περισσότερος διάλογος, περισσότερη συναπόφαση στο μέλλον με το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, κυρίως αν υπάρξει και σχετική τροποποίηση των συνθηκών τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά μας αρχίζουμε να προδικάζουμε τι θα γίνει, διότι συζητάμε στο Ευρωκοινοβούλιο ε, τη δημιουργία κοινοβουλευτικής δομής ούτως ώστε να εκπροσωπούνται οι χώρες της Ευρωζώνης που θα μπορούν να συνομιλούν με σας με, το Eurogroup στο Συμβούλιο. Ποια είναι η υποψή σε αυτή την πρωτοβουλία και τι σχέσεις θα μπορούσαμε να διατηρήσετε στο μέλλον με το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκ. Δεν θα ξαναφερθώ στη θεολογική συζήτηση που αναφέρατε. Ίσως αρκετά υπόθηκαν. Το πρώτο ερώτημά σας ήταν το εξής. Εάν ζητήθηκε άποψη του Επιτρόπου, φαντάζομαι για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αυτό εννοείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα παρούσα και πάντα μας συμβουλεύουν στα διάφορα θέματα και όσον αφορά αν είναι κάτι νομικά εφικτό αν μπορεί κάτι να γίνει στα πλαίσια των παρόντων νόμων και των πλαισίων. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι δεν μας είπαν ότι όχι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ήταν κατά κάτι κατά των συνθήκων ή κατά των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πάντα δίδονται οι σωστές συμβουλές και πάντα κάποιος θα πάρει το λόγο και θα πει «Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται». Άρα πάντα ισχύει αυτό το τεστ, γίνεται για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που αναφέρατε. Είναι διακυβερνητικής φύσεως, είμαι υπέρ του διαλόγου, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ευρεία υποστήριξη τουλάχιστον από πλευράς κρατών μελών για να κινηθούμε προς συναπόφαση σε αυτά τα ζητήματα. Διάλογος, ναι, εγώ είμαι πολύ ανοιχτός όσον αφορά το διάλογο, Είμαι πρόθυμος να έρχομαι στο Κοινοβούλιο και να μιλώ στην Επιτροπή σας για θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup. Είμαι υπέρ, ε, πολύ υπέρ διαλόγου, δηλαδή ε, Επίσης, οι Επιτροπές Εθνικών Κοινοβουλίων και το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετέχουν στην, ε, στα θέματα αυτά στη συζήτηση μακροοικονομικής πολιτικής. Αυτή είναι η απάντησή μου. Καλώς, ευχαριστώ. Μπορούμε να πάμε στο Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Είναι εισηγητής για το ΜΥΦΙΤ, αλλά δεν νομίζω ότι ανακατεύεται εκεί προς με αυτό. Ευχαριστώ, δεν πρόκειται να μιλήσω για το θέμα αυτό. Κύριε Ντάσελμπλουμ, εγώ νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα προέκυψε από δύο πράγματα. Καταρχήν, υπάρχει το πρόβλημα του ότι μετατέθηκε το βάρος όχι στους φορολογούμενους, αλλά στους μικρούς καταθέτες. Και η απόφαση που πήρατε επίσης ε, ομόφωνα είχε σαν, σαν αποτέλεσμα να κυρώσετε το, το σύστημα το τραπεζικό της ε, Κύπρου και είπατε ότι το μοντέλο αυτό το οποίο έχει αυτές τις ε, ιδιαίτερες ε, φορολογικές διευκολύνσεις ότι θα μείνει ακέραιο. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Θέλετε εσείς να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, θα εξασφαλίσετε ότι αυτό το σύστημα που οδήγησε στην κατάρρευση της Κύπρου θα μεταμορφωθεί και ότι η Κύπρος θα μπορέσει να προχωρήσει σε ένα πιο λογικό ε, χρηματοπιστωτικό μοντέλο, όχι μοντέλο πλυντηρίου χρημάτων και υποστήριξη των μεγάλων καταθετών που οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Μιλάτε για μεγάλη απώλεια εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Και δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι η συζήτηση που ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων ότι είχε αρνητικά αποτελέσματα για, τους, ε, για την εμπιστοσύνη των καταθετών. Μετά από μερικές μέρες τώρα μπορώ να πω ότι η συζήτηση ήταν πιο έντονη από ότι η πραγματική αντίδραση των αγορών και των καταθετών. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτό φάνηκε τις τελευταίες μέρες οι αγορές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι έχουμε εμείς ως πολιτικοί και διαμορφωτές της πολιτικής. Από ό,τι νομίζουμε ότι θα έχουν οι αγορές είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη. Η συζήτηση αυτή λοιπόν μας δείχνει ότι θα έπρεπε από την αρχή να είχαμε καλύτερη επικοινωνία για τη διαφορά μεταξύ αυτών που κάνουμε εμείς και του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Εγώ δεν θα μιλούσα όμως για μια μεγάλη απώλεια εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή ανάλυση. Λέτε επίσης ότι το σύστημα, ότι η λύση που προτείνουμε τελικά διατηρεί το επιχειρηματικό μοντέλο της Κύπρου. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε και πολλές από τις συμφωνίες θα, επεξεργα... θα τύχουν επεξεργασίες περισσότερο στο μνημόνιο κατανόησης. Έχουμε μιλήσει για πιο στεναρό έλεγχο της, ε, του ξεπλήματος χρημάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όχι μονάχα για το κατά πόσο οι κανόνες και οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί, έχουν ε, αναθεωρηθεί με συγγνώμη, αλλά και κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά στο πλαίσιο της κρίσης. Έχουμε πολλά λοιπόν πράγματα να πράξουμε. Και δεύτερον, το πρόγραμμα θέλει να επιτύχει και μια αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς και το επιχειρηματικό μοντέλο της Κύπρου. Και τέλος, τρίτον, το αποτέλεσμα τη εφαρμογή αυτού του μοντέλου και του προγράμματο θα είναι μια σημαντική μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Έτσι έχουμε ουσιαστικά τροχοπεδίσει την χρηματοπιστωτική πορεία της Κύπρου. Θέλουμε όλοι να επιτρέψουμε η Κύπρος και ο τομέας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ξαναξεκινήσει σε μικρότερο μέγεθος, σε υγιείς συνθήκες, με λογική φορολογία, και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κατά, της, κατά του ξεπλήματος χρήματος και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Α, μου έχει μείνει ακόμα ένα λεπτό, αν κατάλαβα καλά. Ένα σύντομο ερώτημα. Μπορεί οι αγορές να έχουν καταλάβει αυτό που είπε ο εμείς όμως εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρώπης και όχι τις αγορές. Λένε ότι πληρώνουν, οι πολίτες πληρώνουμε τρεις φορές, πληρώνουμε σαν φορολογούμενοι, πληρώνουμε φορολογία και στους τόκους και τώρα μας καλούν να πληρώσουμε και σαν καταθέτες. Αυτό είναι η κρίση εμπιστοσύνη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Για τις αγορές το ίδιο τους κάνει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους τους απλούς οι οποίοι πληρώνουν την ύφη. Um, well, just... Να πω απλώς ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων στην Κύπρο δεν είναι αποταμιευτές αλλά επενδυτές. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μία απόλυξη σε αυτό το πρόβλημα που να είναι πιο ισοδίκαια. Το είπα στο παρελθόν και ελπίζω ότι η Κύπρος θα θέσει προτάσεις που να ακολουθούν αυτό το οδηγονήμα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τα θέματα αυτά την Παρασκευή το βράδυ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές ότι η εμπιστοσύνη στο, στην εγγύηση μέχρι 100.000 των καταθέσεων είναι απαράγραπτη. Έρχομαι στους τελευταίους ομιλητές. Θα σας δώσω λίγο χρόνο, αλλά σας παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Ο Τις Μπέρμαν από τους σοσιαλιστές και μετά η Ρόδη Κράτσα, προτού ε, δώσει απαντήσεις ο κύριος ε, Ντέισελ Κύριε Ντέσεπλουμ, πολύ χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Ακόμα κι αν μόνο επειδή δείχνετε στους ε, ε, συναδέλφους σας ότι υπάρχει μέλλον μετά, του, μετά τη θέση του βοηθού Ευρωβουλευτή. Αυτό δείχνετε στους συναδέλφους εδώ βοηθούς. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ως ε, πρόεδρος της, του Eurogroup ανησυχείτε για την τεράστια ευθύνη που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια με κάθε κόστος έχει δεσμευθεί να ε, κρατήσει εν ζωή την, ε, την Ευρωζώνη. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει πρωτοβουλίες για να μειώσει την πίεση που δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να βρει άλλον ορισμό της αλληλεγγύης μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ευρωζώνης. Και τι σημαίνει αυτό. Ή ο σημερινός επιμερισμός των κινδύνων μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των χωρών της Ευρωζώνης είναι ε, ε, αρκετό αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, για το πλυντήριο που ανέφερε ο συνάδελφος Βέμπερ προηγουμένως, άλλο είναι το να συμφωνήσουμε ότι η Κύπρο σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, πρέπει να καταπολεμήσει αυτή την πρακτική, όμως όλο αυτό το, το, το ξέπλυμα, η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη για να μην έχουμε μόνο έναν υγιή χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και να υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών υπό αυτή την έννοια. Ευχαριστώ. Κύριε Κατσά. Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, παρότι με Ελληνίδα δεν θα αναφερθώ στο θέμα της Κύπρου, νομίζω ότι συζητήθηκε διεξοδικά θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των ανισοτήτων μεταξύ βορρά και νότου, περιφέρειας και κέντρου, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στην Ευρωζώνη, οι οποίες ε, έχουν αυξηθεί με τις συνέπειες της ε, δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Μας έχει απασχολήσει πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και πρόσφατα είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ντράγκη που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και αναφέρθηκε στην ε, διαφορά παραγωγικότητας και κόστου εργασίας ως βάση αυτής της ανισότητας μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ήθελα να σας να επισημάνω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες ελπίζουμε για ανάκαμψη, επιβαρύνονται από αυτή την ήδη διαφορά που υπάρχει στην Ευρωζώνη ως προς την διάθεση κεφαλαίων και ως προς το κόστος του δανεισμού. Άρα ένας φαύλος κύκλος στην αντιμετώπιση αυτών των διαφορών. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει μια στρατηγική της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, πού βασίζεται αυτή η στρατηγική και θα σας ρωτήσω πώς κρίνεται τα προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης εκεί που εφαρμόζονται στη χώρα μου ζούμε ιδιαίτερα τις συνέπειες ε, αν τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των διαφορών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν πράγματι μεγάλες ε, διαφορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες από αυτές ε, αποτελούν διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου και σίγουρα η κρίση έχει εντείνει αυτές τις διαφορές. Ε, η παρατήρηση που έκανε ο Μαριό Ντράγκη ήταν ότι προκειμένου η Ευρωζώνη στο σύνολό της να καταστεί πιο ανταγωνιστική, θα πρέπει και εμείς να γίνουμε πιο καινοτόμοι, να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να μειώσουμε το εργατικό κόστος ε, και τον λόγο του σε σχέση με την ε, παραγωγικότητα. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα των χωρών του Νότου ή του Βορρά. Νομίζω ότι είναι ζήτημα για όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, και για τις χώρες ε, της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά και στις κάτω χώρες είναι θέμα αυτό. Δεύτερον, πολλά από τα προγράμματα που ήταν απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης σε ορισμένες χώρες συνέβαλαν και σε αυτό το, στοιχείο ε, του εργατικού κόστους και της παραγωγικότητας. Αν εξετάσουμε λοιπόν το εργατικό κόστος σε χώρες της Νότιας Ευρώπης αυτή τη στιγμή, η παραγωγικότητά τους αυξάνεται ταχύτατα. Και η σχετική τους θέση σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται εργοστάσια μεταφέρονται από τον Βορρά στον Νότο. Βεβαίω οι άνθρωποι στον Βορρά δεν ε, χαίρονται, αλλά πράγματι υπάρχουν εργοστάσια που μεταφέρονται στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Και αυτό συνδέεται με τι μεταρρυθμίσει που έχουν πραγματοποιηθεί. Όμω ε, το βασικό είναι ότι κάποιε φορέ ε, η κουβέντα είναι για το αν θα πρέπει ο Βορρά να είναι λιγότερο ανταγωνιστικό, να εξάγει λιγότερα για να αναπτυχθεί ο Νότο για μένα θα έπρεπε ολόκληρη η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ομάδα από διεθνή σκοπιάς να γίνει ε, ισχυρότερη. Να εξάγουμε περισσότερα ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί αν μόνο επικεντρωθούμε στην ισορροπία μεταξύ, ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσουμε πολλές ευκαιρίες στο διεθνές εμπόριο. Και αυτή τη στιγμή οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης βρίσκονται εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλες περιοχές του κόσμου που υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Και αν εμείς ε, όλες μαζί οι χώρες ε, μπορούμε να ε, συμμετάσχουμε σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη και αυξήσουμε τις εξαγωγικές μας δραστηριότητε ε, εκτός, τότε μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, είναι ο ένας χάνει, ο άλλος κερδίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, συγγνώμη, αγαπητέ συγγνώμη που ξέχασα να απαντήσω στη δική σου ερώτηση. Είμαι και ο πρώτος και ο μόνος που θα σε συγχωρήσει αυτομάτως. Uh, Με ρώτησε για την ε, ευθύνη ε, που αναλαμβάνει η ΕΚΤ και μήπως είναι υπερβολικά μεγάλη αυτή η ευθύνη. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι αναπόφευκτο. Όμως σε, σε μια υγιή και βιώσιμη κατάσταση μετά την κρίση, βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα προγράμματά της θα πρέπει να μειωθούν σε εύρος και διάσταση. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίως και το αναγνωρίζει αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ε, αναπόφευκτα λοιπόν η ΕΚΤ θα διαδραματίσει αυτό τον σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερα επικοδομητικό μάλιστα. Προς το παρόν λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι από πλευράς ε, ε, φορέων χάλαξη πολιτική ε, και θεσμικών οργάνων και κρατών μελών έχουμε καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή μα για το μέλλον. Το δεύτερο ερώτημά σου αφού αφορούσε την φόρο διαφυγή και το ξέπλυμα χρήματο. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης για όλες τις χώρες είναι η συνεργασία μεταξύ μας γιατί είναι ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Ε, τα φορολογικά συστήματα είναι ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τα φορολογικά συστήματα, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε από κοινού. Είναι η μόνη λύση. Αυτό είναι μάλλον ένα ερώτημα προς ε, τον ε, Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών. Το ξέρω και προσπαθώ να είμαι όσο πιο ανοιχτό και ειλικρινής η μόνη λύση είναι να γίνει αυτό διεθνώ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Σόφι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ως ε, εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων, ε, να σας εγχαρώ ε, και να σας καλωσορίσω. Ελπίζουμε να σας δούμε πολλές φορές στο μέλλον. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν για την Κύπρο σήμερα. Όμως υπάρχουν και φήμες ε, στα ΜΜΕ και για άλλες χώρες με συστημικό κίνδυνο που θα μπορούσαν να έρθουν στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι και εσείς δεν θέλετε να εκφέρετε γνώμη, αλλά είμαι, έχω μια περιέργεια. Δεύτερον, είπατε σωστά ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές. Ωστόσο, διαπιστώνω ότι παρά το έκτακτο της κατάστασης, το κρίσιμο της κατάστασης, ε, ακόμα οι εθνικές ε, κυβερνήσεις ασχολούνται με το εθνικό τους, ε, τους εθνικούς τους ψηφοφόρους και το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε μονίμως σε μια κατάσταση διαχείρισης κρίσεων παρά χάραξης πολιτικής για το μέλλον. Αναφερθήκατε στη συμπλήρωση της εργαλειοθήκης ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αναγκάσετε τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και τέλος, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φήμες για ε, τελεσίγραφο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε ό,τι αφορά και την Κύπρο θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας θέση από αυτού. Ευχαριστώ κυρία Νετφέλτ για τις ερωτήσεις σας. Το πρώτο ερώτημά σας αφορούσε τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσουν ε, πρόβλημα αν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Δεν μπορώ να σε αυτό. Εν γέννη, η Ευρωζώνη διέρχεται μια περίοδο μεγαλύτερης ε, σταθερότητας και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να εργαστούμε για όλα τα μέσα, για όλους τους μηχανισμούς που χρειαζόμαστε για καλύτερη, καλύτερη συντονισμένη μακροοικονομική πολιτική. Δεν θα αναφερθώ για μελλοντικούς ενδεχόμενους κινδύνους. Ζητήσατε ευρωπαϊκές λύσεις και εγώ το ίδιο, απευθύνεται έκκληση και οι εθνικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να εστιάζονται πολύ στο εκλογικό τους σώμα αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα. Παραφράζω αυτά που είπατε. Ε, για πολιτικούς, εθνικούς ή ευρωπαίους πρέπει πάντα να βρίσκουν τρόπους για να εφαρμόζουν αυτό που είναι σωστό και αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει μαζί να παρασύρεις και το εκλογικό σου σώμα. Ε, να συμφωνεί. Διαφορετικά θα έχει πολύ σύντομη θητεία και αυτό που έθεσα στόχο δεν θα είναι βιώσιμο αυτό που θες να κάνεις διότι οι επόμενοι πολιτικοί θα αλλάξουν την πορεία σου εντελώς. Οπότε πάντα υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σε αυτά που κάνουμε, πώς μπορούμε να έχουμε συμπαραστάτες τους ψηφοφόρους μας, τους λαούς μας. Και καμιά φορά προχωρώντας κανείς πολύ γρήγορα, ε, χαλάς τη τάξη τη παρέλαση του ΣΥΠΗΝ. Πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και να έρχονται και άλλοι μαζί σου. Ε, και έχουμε και τα θέματα τη Τραπεζική Ένωση. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, καμιά φορά θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα. Από την άλλη, αφετηρία της όλης, του όλου προγράμματο στην Τραπεζική Ένωση, που είναι από τα μεγαλύτερα προγράμματα στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση, ήταν μόλι πριν από ένα εξάμεινο. Και ήδη ε, το Δεκέμβριο συμφωνήσαμε εντό του ΕΚΟΦΗΝ στο πρώτο οικοδομικό στοιχείο αυτή τη Τραπεζιτικής Ένωση. Α μην αλληλοκατηγορούμαστε. Το έργο που γίνεται για την Τραπεζική Ένωση προχωρά αρκετά γρήγορα και θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και Σόφη σα ρώτησε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Α, και κάτι άλλο να, βάλω, να προσθέσω κι εγώ, οπότε να απαντήσετε γενικά για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούσαμε ότι κατά έργα των συνομιλιών υπήρξε απειλή απόσυρσης της ε, ρευστότητας ανάγκης και όταν φαινόταν ότι χρειαζόταν κάποιος χρόνος ε, και όταν φαινόταν ότι κάτι μπορούσε να γίνει έμενε ε, η ρευστότητα όσο χρειαζόταν τελικά. Και όπως είπε η Σόφη, ίσως ε, από τη Δευτέρα να αποσυρθεί, να σταματήσει αυτή η ρευστότητα. Ποια είναι η άποψή σας δηλαδή της χρήσεως ε, για την ε, ρευστότητα ανάγκης που μία χορηγείται, μία αποσύρεται, ε, γίνεται αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απειλεί. Νομίζω ότι κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο μέσα στα πλαίσια της εντολής τους και η ELA, δηλαδή η έκτακτη παροχή ρευστότητος, μπορεί να δίδεται σε αυτές τις τράπεζες και μόνο που είναι φερέγγες και αν είναι πράγματι σε δυσκολία μια τράπεζα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια προοπτική στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ένα πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης ώστε αυτές οι τράπεζες να βρεθούν σε ασφαλείς λιμένες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρά μέσα στα πλαίσια της εντολής της και είναι ανεξάρτητη. Αυτοί πρέπει να κρίνουν αν μπορούν να συνεχίσουν με την παροχή της έκτακτης υποστήριξης λεπτότητος και από ό,τι κατανοώ θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κατεπήγον να βρεθεί ένα πρόγραμμα για τη διάσωση των τραπεζών και μπορούν να υποστηρίξουν με την έκτακτη παροχή ρηστότητος εάν υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό καταδεικνύει λοιπόν πόσο κατεπήγον είναι το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατό. Και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος, όπως είπα και στην αρχή. Ήταν δύσκολη η πρώτη σας ε, ε, παρουσία ενώπιον της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε που παραμείνατε πιστός στις θέσεις σας και ελπίζουμε ότι και στις επόμενες επαφές μας προβλέπετε να ξαναβρεθούμε το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο κύριος Ντέισελ Μπλόμ. Πάμε στις ψηφοφορίες. Ένα-δύο λεπτά διακοπή ώστε να μπορέσουν να έχουν όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας και να φύγουν αυτοί που θέλουν να φύγουν. Okay, we, we do... Καλώς, πρέπει να ψηφίσουμε, πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, καθίστε. Okay, thank, thank, thank you very much. Um, right, well, the first, the first matter... Το πρώτο θέμα είναι το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Στατιστικά Στοιχεία και ο διορισμός του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ετέθη όταν αυτή η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Στατιστικά Στοιχεία συστάθηκε στην προηγούμενη θητεία. Ήμουνα η πρώτη από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου ακολουθήθηκε από τον Έντουαρτ Σεκλούνα που είναι τώρα υπουργός οπότε είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η θέση αλλά Λίαμ Νουαγκόγκ είναι ο υποψήφιο. μόνο έναν έχουμε μόνο έναν υποψήφιο προτείνω λοιπόν διαβοή να εγκρίνουμε αυτή την υποψηφιότητα And watch out where you're going. και πρόσεξε που πας μετά Λιάμ αν θες να πάει στο λόγο πολύ σύντομα, έχεις το λόγο. Απλώς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι σημαντική, διότι πρέπει το Κοινοβούλιο να μπορεί να επαγρυπνεί όσον αφορά την ποιότητα και την εξοπιστία των στατιστικών στοιχείων. Είναι πρωταρχική σημασία για μια καλή μακροοικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Εν ονόματί σας λοιπόν θα φροντίσω γι' αυτό ακριβώς, να εργαστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που μπορεί να μάθει κανείς για τα όσα συμβαίνουν όταν παρίσταται στις συνεδριάσεις. Το ξέρω από τη δική μου εμπειρία. Προχωράμε στο σημείο 12 την ψηφοφορία όσον αφορά το usage. Μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε πώς λειτουργούν οι κάρτες, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία με τις κάρτες για να ξέρουμε τι γίνεται. Πατήστε τα κουμπάκια σας. Το κουμπάκι της χαράς. Καλώς. Ένας είναι συνδεδεμένος αλλά δεν ψηφίζει. Φαντάζομαι ότι είναι σκόπιμο αυτό. 29 ικανοποιημένοι, ένας μη ικανοποιημένος, 8 δεν γνωρίζουν. Οπότε... Ζαν Πολ, ο κύριος Γκοζές, δεν έχεις κάρτα. Να προσθέσουμε άλλον έναν λοιπόν. Πρέπει όμως να μας δείχνετε τι ψηφίζετε. Υπάρχει άλλος που δεν έχει την κάρτα του. Όχι. Μόνο ένας άτακτος συντονιστής. Δεν νομίζω ότι δουλεύει η πιστοτική, Ζαν Πολ, σε αυτή τη σχισμή. Επιτροπή Οικονομικών. Μπορεί να αγοράσετε ψήφο. Όχι, όχι, συγγνώμη. Αστείευομαι. Λοιπόν, ας, αρχίσουμε. Τέλος πάντων, ας ψηφίσουμε. Η πρώτη αφορά τις αμοιβέ σχετικό θέμα, συμβιβαστική α, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές το πρώτο τμήμα εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι άλλους δύο ένας να ψηφίσει ακόμα ψηφίσαν όλοι πέρα ψηφοφορίας 22 με 16 εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Πάμε στην τροπολογία 9. Όχι. Στη συμβαστική Β. Okay, compromise B. although. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική C λατινικού υπέρ. Α, είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται. 17 υπέρ, 22 ψήφοι εναντίον. Συμβιβαστική D, συμβιβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε άμα τη βρω, τροπολογία 22, τροπολογία 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ή e, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα ελέγξουμε Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όπως θα ανέμενε κανείς από μια συμβαστική τροπολογία. Συμβιβαστική F. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ας ελέγξουμε όπως κάναμε και πριν ψήφισαν όλοι άλλος ένας πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 23 ψήφους ε, εναντίον 17 υπέρ πάμε σε προφορική τροπολογία δική μου της Προέδρου να συμπεριληφθεί η συνθισμένη διατύπωση που αφορά τους πίνακες συσχετισμών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε για την τροπολογία 8 έλεγχος τροπολογία 8 έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 21 18 19 21 19 ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, συμβαίνοντας τον Ζαν Πολ, 5 ψήφοι κατά και 5 αποχές. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Το ίδιο 30 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 5 εποχές. Πρέπει ε, ο εισηγητής ε, επιθυμεί να κάνει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Όπως συνηθίζεται, στα πλαίσια των κανονικών διαδικασιών, επειδή δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, αν κάποιο στην Επιτροπή θέλει να πάει στην Ολομέλεια, μπορώ να πάω στην Ολομέλεια. Αν υπάρχει ομοφωνία να πάμε αμέσω στο Συμβούλιο, να πάμε στο Συμβούλιο. Εγώ θέλω να είμαι πολύ δίκαιο, το συζητήσαμε εκ των προτέρων. Παρόλο που η πλειοψηφία στο τέλο ήταν πολύ μεγάλη. Το αφήνω στου συναδέλφου. Αν θέλετε να πάμε στην Ολομέλεια, να πάμε. Διότι το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει ακόμα Οπότε από πλευράς δημοκρατικής υπάρχει ακόμα χρόνος. Ναι, μου λένε εδώ ότι η Ιρλανδική Προεδρία σαν σημείωμα θα ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο τον ε, Απρίλιο προσπαθώντας να πετύχει μια γενική προσέγγιση. Οπότε το ερώτημα είναι θέλουμε να το θέσουμε αυτό στην Ολομέλεια μαζί με δεχόμενες ε, αλλαγές θα μας έδινε περισσότερο χρόνο ίσως για να κάνουμε τελευταίες μικρορυθμίσεις αν ήταν απαραίτητο. Διερωτώ αν, αν το ζητήσει ένας ή η πρόεδρος μου πάμε στην Ολομέλεια και εγώ είμαι έτοιμο ε, να συνεργαστώ με τους σκιώδεις και να βρούμε λύσεις για τα πάντα. Ε, όπως είχαμε και λύσεις μέχρι πριν από μερικές ε, μέρες. Οπότε εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Αν ένας ζητήσει να πάμε στην Ολομέλεια, ξεκάθαρα το λέω ξεκάθαρα, θα το κάνουμε. Η Πρόεδρος. Ο Γουλφ το πρότεινε. Λοιπόν, έτσι έχουμε και μερικές μικρορυθμίσεις ε, να κάνουμε, άρα ίσως χρειαστεί να πάμε στην Ολομέλεια. Οπότε το θέτουμε στην Ολομέλεια. Πάμε στην Ολομέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, αλλά ας δούμε τι θα γίνει στην ε, Ολομέλεια. Καλώς. Πάμε Στο 13 η κοιτοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου βοήθειας που χορηγείται στα κράτη-μέλη που δεν έχουν το ευρώ σαν νόμισμα είναι η έκθεση της Ντανούτα Χούμπνερ. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, το αρχικό κείμενο δεν ψηφίσαμε. Α, το αρχικό κείμενο στην παράγραφο 2, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε όμως. Γιατί ήμουν αφηρημένη. Για να μην ειλικρινείς κιόλας. Πέρας. Και υπεραπορρίπτεται, ναι. Τροπολογία 19. Υπερ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπερ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο για την παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική F. Ναι, ναι. Συμβαστική F λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το αρχικό κείμενο στην παραφό 5 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Πάλι το, η τρίτη παύλα στην παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική I σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο στην δέκατη παύλα υπέρ κατά αποχές δεκτό 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή πέμπτη παύλα στην παραγωγό 5 υπέρ κατά αποχές δεκτό δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο τροπολογία 57 υπέρ κατά δεκτή, συμβαστική και υπέρ κατά δεκτή. Το αρχικό κείμενο της παράγραφου 6 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Αιτιολογική σκέψη. Μπορούμε να τις πάρουμε όλες μαζί τις αιτιολογικές σκέψεις. Όλες μέχρι την αιτιολογική σκέψη Β, αιτιολογικές αναφορές και αιτιολογική σκέψη Β, πάμε υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Κάναμε την αιτιολογική σκέψη Σ ή όχι. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2. Υπέρ κατά δεκτή, 3, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά δεκτή, 5 υπέρ Δεν ψηφίσαμε την τροπολογία 3, λέει η κυρία Φερέιρα. Εντάξει, έχετε δίκιο. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή αιτιολογική σκέψη F, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, απορρίπτεται συγγνώμη, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή, το συνολικό κείμενο λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Ένας ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Κλείνω την ψηφοφορία. 35 εναντίον μιας, 36 μαζί με τον Ζαν μία κατά και τρεις αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φοβάμαι ότι πρέπει να σας πω ότι τελειώσαμε και η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 26 Μαρτίου στις 9 το πρωί και στις 3 η ώρα επίσης, στις 26. Δεν έχουμε τίποτα την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχω ακόμα αποφασίσει την επίσημη ακύρωση της συνεδρίασης. Ίσως για λόγους σοφροσύνης πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να συνεδριάσουμε εάν υπάρξει πρόβλημα. Θα σας ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατό. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 11 Απριλίου 9 έως 12. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει για να σας πω αν θα ακυρωθεί ή όχι η συνεδρίασή μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.